thank you very much everybody. Welcome. Ωραία. Καλώς ήρθατε στο τμήμα ΕΚΟΝ της Επιτροπής Οικονομικών και Νοσματικών Επιθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το διάλογο που διεξάγουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την συμβολή σας που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον εκδημοκρατισμό του εξαμήνου. Με το εξάμεινο η διαδικασία καθορισμού των προτεραιοτήτων έχει αλλάξει. Ορισμένα κράτη-μέλη, πολλά κράτη-μέλη βλέπουν την ε, Ευρώπη να παρεμβαίνει ε, στην οικονομική της πολιτική και μάλιστα στις χώρες που υπάγονται σε προγράμματα πολλές από τις απαιτήσει ε, σχεδόν επιβάλλονται στις εθνικές αρχές παράλληλα να γνωρίζουμε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα τουλάχιστον όσον αφορά την λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ένωσης. Στην ουσία είναι διακυβερνητικές αποφάσεις ε, και κλεισμένων των θυρών με βάση συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιος τελικά αποφασίζει τους στόχους πολιτικής και ποιος φέρει την ευθύνη για αυτούς. Τώρα λοιπόν θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ελπίζω συζήτηση για τον τρόπο ανοίγματο και εκδημοκρατισμού αυτών των διαδικασιών. Καλωσορίζω τον Ντόμινικ Χάνικεν, που είναι επικεφαλής της Κοινής Επιτροπής για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, τον Γκούντρουν Γουλφ, που είναι αναπληρωτής, διευθυντής της ε, ομάδας μελετών ε, που βασίζεται στις Βρυξέλλες Λιδεμπρούγκελ και τον κύριο Κολινιό, που είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών στην ε, Σχολή ανωτέρων πολιτικών ε, σπουδών στην Πίζα που λέγεται Αγία Αρνή. Πρώτα θα ακούσουμε τον καθηγητή Κολινιόν. Έχει αλλάξει επανειλημμένα σειρά, αλλά συμφωνήσαμε με τους ομιλητές ότι με αυτή τη σειρά θα πάρουν το λόγο. Ο καθένας θα κάνει μια παρουσίαση 10 λεπτών και μετά αν υπάρχει χρόνος φυσικά θα λάβετε το λόγο κι εσείς σας παρακαλώ λοιπόν να συμπληρώσετε ε, τα έντυπα για τους ομιλητές όπως και σήμερα το πρωί. Και στόχος μας θα είναι να ομιλούν κατά σειρά δύο εθνικοί βουλευτές και ένας ευρωβουλευτής. Αλλά ανάλογα με τις αιτήσει μπορεί να ποικίλει η εναλλαγή των ομιλητών. Σας καλωσορίζω. Κούντρουμ, μπορείτε να ξεκινήσετε. Εκεί θα έχετε το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, αξιόλογοι εθνικοί και ευρωβουλευτές, εθνικοί βουλευτές και βουλευτές του Ευρωβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω δυνατότητα να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τη Δημοκρατία. Πρώτα, να παρουσιάσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και μετά, για λίγο, θα συζητήσουμε για τις ε, λύσεις που έχουν ε, τεθεί σε εφαρμογή και να δούμε ποια είναι τα όρια αυτών των λύσεων από πλευρά νομιμοποίησης και περαιτέρω εξελίξεων στην ε, ε, οικονομική πολιτική και στον οικονομικό συντονισμό στην Ένωση. Πρώτον, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι χώρες της ζώνης ευρώ έχουν μειωμένη κυριαρχία. Τι εννοώ. Οι χώρες αυτές έχουν ε, πολύ περιορισμένη κυριαρχία για μια σειρά τομείς. Δεν έχουν ε, κυριαρχία για την νομισματική πολιτική. Σαφές αυτό. Αλλά δεν είναι απλώς ο τομέας της ε, νομισματικής πολιτικής. Έχει να κάνει και με την φορολογική ή δημοσιονομική πολιτική υπάρχουν ε, δύο όρια που είναι καταφανή. Πρώτο το όριο που επιβάλλουν οι χρηματαγορές για την ε, δυνατότητα πώλησης ομολόγων. Βλέπουμε ότι διάφορες χώρες μέλη έχουν δυσκολίες ε, στην πώληση των ομολόγων τους. Άρα περιορισμός της κυριαρχίας. Περιορισμό του καθορισμού των ελλημάτων που θα ήθελαν να έχουν, γιατί υφίστανται υψηλέ πιέσει από τις αγορές. Πρώτο όριο, το οποίο διαπιστώνουμε. Και δεύτερο, που σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες εκτός Ευρωζώνης που έχουν πολύ περισσότερη δυνατότητα να πολλούν ομόλογα και υφίστανται πολύ λιγότερε πιέσει από τι ε, χρηματαγορές. Άρα έχει χαθεί για μεγάλα τμήματα τη Ευρωζώνης η δημοσιονομική κυριαρχία. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη συμμερίζονται υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες. Που είναι πιο συγκεκριμένα στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά πρόσφατα εξαπλώθηκαν και στους ε, τομείς της μη δημοσιονομικής πολιτικής. Άρα αυτός ο συνδυασμός πιέσεων από τη συνθήκη και τις αγορές περιορίζει την κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Και πώς θα αντιμετωπιστεί το οικονομικό πρόβλημα καθώς και το πρόβλημα νομιμοποίησης που προκύπτει από τις ε, συγκεκριμένες αυτές καταστάσεις. Τι προτείνεται αυτή τη στιγμή ως επίλυση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, δεν θυμάμαι τώρα τι σημαίνουν ε, τα διάφορα αρχικά, η συνθήκη για την σταθερότητα και την ε, διακυβέρνηση της ΟΝΕ, βέβαια δεν είναι μόνο για δημοσιονομική για τον ε, συντονισμό της δημοσιονομικής αλλά και γενικά της οικονομικής πολιτικής. Επίσης τώρα έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Διακυβερνητικό σώμα που έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει ενίσχυση στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και αυτή τη στιγμή είναι μόνο στα κράτη-μέλη, όχι στις τράπεζες. θα ήταν ένα βήμα περαιτέρω να μπορεί να διασώζονται απευθείας τράπεζες. Αυτό σε ορισμένα κράτη-μέλη θα προϋπέθεται τροποποίηση της νομοθεσίας. Τώρα, η νομοποίηση αυτών των ρυθμίσεων απορρέει από αποφάσεις ή μάλλον καλύτερα πρώτα απ' όλα από το ότι είναι συνθήκη που έχει υπογραφεί από κυρίαρχα κράτη-μέλη που συμφώνησαν λοιπόν να τηρούν κάποιους κανόνες και αμεσότερα οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου λαμβάνονται από το Συμβούλιο που αποφασίζει πότε κάποιο έλλειμμα είναι υπερβολικό, αλλά παίζει και κύριο ρόλο για τις διαδικασίες, για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και για θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την μακροοικονομική πολιτική στο μέτρο που δεν είναι δημοσιονομική. Λοιπόν, πολύ ευρύς τομέας αρμοδιοτήτων. Τώρα, Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αγωνιστεί σκληρά για να αυξηθεί η κοινοβουλευτική νομιμοποίηση. Όμως ε, η βάση από τις συνθήκες είναι περιορισμένη για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, διότι σύμφωνα με τη συνθήκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατακτήσει το μέγιστο εφικτό των ε, αρμοδιοτήτων του. Επίσης υπάρχει ένας διάλογος που επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ζητήσει απολογισμό από τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, αλλά ακόμη και από υπουργούς ε, εθνικών κυβερνήσεων, να τους καλέσει, να παρουσιάσουν την πολιτική τους και να κάνουν έναν απολογισμό. Αυτή είναι οι πυλώνες της νομιμοποίησης. Είναι δηλαδή στην ουσία δυνατότητες επηρεασμού της πολιτικής πριν αποφασίσει το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο προσπαθεί να συμμετάσχει και στην ετήσια μελέτη για την ανάπτυξη και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υπόλοιποι μηχανισμοί, αλλά στην ουσία το Συμβούλιο και η Επιτροπή παίζουν τον πρώτο ρόλο στον καθορισμό της λειτουργίας αυτών των μηχανισμών. Το θέμα λοιπόν της ε, νομιμοποίησης είναι στην καρδιά της αποτελεσματικότητας όλης αυτής της διαδικασίας. Κάναμε μία μελέτη προσπαθώντας να δούμε σε τι βαθμό τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν στις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και διαπιστώσαμε ότι μετά την διατύπωση των συστάσεων περιορισμένη είναι η δυνατότητα συζήτησης των Εθνικών Κοινοβουλίων τα οποία δεν συμμετέχουν πλήρως. Πικίλια από χώρα σε χώρα αλλά δεν είναι το απόλυτο πλήρες επίπεδο νομιμοποίησης που θα μπορούσαν να παράσχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είπα λοιπόν ότι νομιμοποίηση ίσον αποτελεσματικότητα. Γιατί μόνοι όσοι έχουν την τελική αρμοδιότητα λήψη αποφάσεων, δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια για του εθνικού προπολογισμού, μόνο τότε, ανεπισμένα δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια, τότε η εφαρμογή της πολιτικής θα είναι αποδοτική. Οπότε, Είμαστε ανάμεσα σε δύο καρέκλες. Έχουμε τρεις επιλογές. Και πρέπει να τελειώνω, το βλέπω. Δηλαδή, τι διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτή την αίθουσα. Οι εθνικοί βουλευτές να έρχονται στις Βρυξέλλες για να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης Καλό θα ήταν αρχικά να υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση. Δημιουργούμε δυνατότητα διαλόγου και διεθνική κοινοβουλευτική συνεργασία. Αλλά το μεγάλο είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμμετάσχουν πολύ περιορισμένα. Δηλαδή οι τρεις-τέσσερις που έρχονται πρέπει να φέρουν την ευθύνη να εξηγήσουν μετά στου 300-500 συναδέλφου τους ποιες αποφάσεις λήφθηκαν και ποιε όχι και γιατί. Άλλη επιλογή. Οι Βρυξέλλες ε, να ε, πάνε σε εθνικές πρωτεύουσες, θα το πω έτσι προκλητικά. Έχουμε δει μερικά τέτοια παραδείγματα. Κάποιοι λοιπόν από την Ευρωπαϊκή... Ο Μάριο Ντράγκη που πήγε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο στο Βερολίνο, πολύ καλό παράδειγμα ενό ευρωπαϊκού θεσμού απευθεία να εξηγεί στου εθνικούς νομοθέτες την πολιτική του αυξάνοντας έτσι την συνειδητοποίηση σε εθνικό επίπεδο του τι συμβαίνει και θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν μαζί του. Επίσης και οι επίτροποι μπορούν να πάνε στα εθνικά κοινοβούλια. Και τρίτη προσέγγιση, και σε αυτήν πρέπει να καταλήξουμε στο τέλος και νομίζω ότι και ο Στέφαν θα συνεχίσει την γραμμή μου, είναι να υπερβούμε τις υπάρχουσες συνθήκες, να αρχίσουμε σοβαρά να εξετάζουμε τι σημαίνει περιορισμένη εθνική κυριαρχία και να συμφωνήσουμε σε ε, από κοινού άσκηση και της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων. Από κοινού άσκηση της νομιμοποίησης. Τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, ούτως ώστε να υπάρξει ένα, μια νέου είδου νομιμοποίηση. Είναι σαφές ότι η διακυβερνητική προσέγγιση έχει σαφή όρια. Πρέπει να περάσουμε τελικά, ας το πω έτσι, μια πιο ομοσπονδιακή εναλλακτική λύση Κάτι που θα σημαίνει να λαμβάνονται ουσιώδεις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φορολογικού τύπου αποφάσεις. Αυτή είναι η ζωτική, η ζωτική ε, εξουσία όπου θα παιχτεί το θέμα της Ευρώπης. Και το θέμα είναι τι ε, κοινοβούλιο μπορεί να έχει τέτοιες δυνατότητε επιβολής φόρων ε, θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Στέφαν Κολινιό είναι ο επόμενος ομιλητής. Στέφαν. Ευχαριστώ Σάρον, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Το ερώτημα που μου τέθηκε είναι ποιος θέτει το θέμα, το θεματολόγιο, την ατζέντα. Ας δούμε λίγο τη θεωρία των αποφάσεων, δηλαδή πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρητικά. Ανά πάσα στιγμή τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να θέλει να πάρει την απόφαση, ε, κοιτάζει την κατάσταση, πώς έχει εκείνη τη στιγμή. Εν συνεχεία, έχει στη διάθεσή του μία δέσμη δράσεων και λαμβάνει υπόψη του τα θετικά της κάθε μίας και τα αρνητικά φυσικά. Η πολιτική είναι να δώσουμε σε αυτόν που λαμβάνει την απόφαση μια συνταχή, ούτω ώστε να επιλέξει τις δράσεις του. Χρειαζόμαστε δηλαδή το άτομο που παίρνει την απόφαση και χρειαζόμαστε και κάποιες ε, συνταγές με βάση τις οποίες θα επιλέξει κάποιες δράσεις αυτό το άτομο. Αυτό στο δημόσιο τομέα σημαίνει όμως και νομιμοποίηση μιας πολιτικής που απορρέει από την αποδοχή της απόφασης, η οποία εξαρτάται από τη διανομή των ωφελών. Εξαρτάται δηλαδή από το πώς αντιδρούν αυτοί που επηρεάζονται από τις ε, δράσεις αυτές. Πώς αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσει τη ζωή τους και τον κόσμο. Αυτός ο ορισμός της νομιμοποίησης που, που σας έδωσα περνάει είναι ένα στάδιο πιο μετά από τον ορισμό της νομιμοποίησης που σας έδωσε ο Γκούντραμ και αφορά την βιωσιμότητα οποιοδήποτε θεσμών και εν προκειμένου των ευρωπαϊκών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Δεν είναι ένας φορέας. Έχουμε συλλογική λήψη των αποφάσεων και μέσα από μια διαδικασία λαμβάνεται συλλογικά μια απόφαση. Το σύστημα το οποίο παράγει αυτές τις αποφάσεις είναι η διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα, είναι πολύ περίπλοκη γιατί υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου, μεταξύ φορέων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ κέντρων αποφώσεις, λήψης απόφασης. Τελικά θα πρέπει να εκφράζονται τα συμφέροντα των εκλογέων τα εθνικά κοινοβούλια αντλούν την νομιμότητά τους από τους ε, ανθρώπους που ψηφίζουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό, αυτό είναι ο λίθο λήθος της ε, δημοκρατικής νομιμότητας. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, δηλαδή η συνταγή για δράση, διατυπώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό γίνεται με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν που είναι συνεταίροι σε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία, συνεχεία, προχωράει ε, στα εθνικά κοινοβούλια και τα εμπλέκει, γιατί εκεί εφαρμόζονται οι αποφάσεις. Και εκεί επηρεάζεται και ο κόσμος από αυτές τις αποφάσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους. Η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων ξεπερνάει το κρατικό επίπεδο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας φορέας, ένας παράγοντας που λαμβάνει τις αποφάσεις. Το ερώτημα τίθεται λοιπόν το ποιο δίνει την νομιμότητα στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Χωρίς ένα, ένα συγκεκριμένο φορέα που αποφασίζει, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει λογοδοσία, να υπάρξει απολογισμός. Είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, να καταλάβουμε γιατί κάποιες αποφάσεις είναι αποδεκτές από αυτούς που επηρεάζονται από αυτές τις αποφάσεις και γιατί κάποιες άλλες όχι. Αυτό το σύστημα πολλαπλής διακυβέρνησης που σας περιέγραψα λειτουργεί εφόσον υπάρχει μια κοινωνική συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνταγές αυτές πολιτικής. στην αρχικές φάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης περί αυτού επρόκειτο. που θα δημιουργηθούν συνεργασίες, συνέργειες, κοινά ωφέλη, οικονομίες κλίμακας. Ποιο είναι το κόστος της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Όλα αυτά τα επιχειρήματα που μας έλεγαν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και η νομιμοποίηση υποστηριζόταν από την αποδοχή από όλους. Όλοι έβγαιναν κερδισμένοι και κανένας δεν έχανε από την ιστορία. Σήμερα όμως, και αυτό είναι συνέπεια σε μεγάλο βαθμό της, της νομισματικής ολοκλήρωσης, τώρα έχουμε πια νικητές και ιτημένους. Δεν φτάνουμε πια σε αυτό το optimum όπου όλοι κερδίζουν. Στη θεωρία της απόφασης η στρατηγική υποκαθιστά τις ε, δυνατότητες. Δηλαδή οι αποφάσεις μου θα ωφελήσουν εμένα μεν, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν μειονέκτημα για κάποιον άλλον και αντιστρόφως. Και επομένως υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Και επομένως σε αυτή τη διαδικασία έχουμε τους ε, νικητές και τους ιτημένους. Ε, Πρόβλημα με την νομιμότητα είναι γιατί οι ιτημένοι θα πρέπει να δεχτούν κάποιες αποφάσεις εάν από την εφαρμογή τους προκύπτουν κάποιες ζημίες, κάποιες απώλειες. Η απάντηση που δίνει η θεωρία μας είναι ότι στην δημοκρατία μπορούμε να δεχθούμε κάποιες ζημίες γιατί υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της πολιτικής, στο μέλλον φυσικά. Η αλλαγή της κοινή γνώμης οδηγεί σε αλλαγή των πολιτικών και εφόσον αυτό το σύστημα παραμένει αξιόπιστο, υπάρχει νομιμοποίηση αυτού του τρόπου λήψης των αποφάσεων. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επειδή έχουμε αυτή την πολλαπλή περίπλοκη διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη, δεν έχουμε τη δυνατότητα ή μειώνεται η δυνατότητα για αλλαγή. Η συνένεση δεν προκύπτει από τη συζήτηση στο λαό, αλλά η συνένεση επιτυγχάνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προκύπτει από συζητήσεις πολιτικής που είναι εθνικές και όχι ευρωπαϊκές. Όταν κοιτάτε την δημοκρατική νομιμότητα πίσω από τις ε, εθνικές εκλογές, θα καταλάβετε ότι είναι ε, περιφερειακές εκλογές. Αλλάζουμε δηλαδή τις εθνικές εκλογές, αλλά ποτέ δεν έχουμε βουλευτικές εκλογές όπου συζητούνται και αποφασίζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι επηρεάζονται από αυτές τις αποφάσεις να μπορούν να εκφράζουν τις αποφάσεις τους. Δεν μπορούν να τις εκφράζουν. Έχουμε λοιπόν αυτή την, αυτούς τους νικητές και νικημένους. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο απονομιμοποίησης της λήψης των αποφάσεων. Και αυτό έγκυται στην καρδιά της ε, κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος δεν πιστεύει πια ότι μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές ε, μέσω των βουλευτικών εκλογών και επομένω τελικά θα απορρίψει το όλο σύστημα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και προωθούνται κάποιες πολιτικές. Καταρχάς υπάρχουν εναλλακτικέ πολιτικής. Αυτό που υπάρχει ε, στην Ευρώπη είναι η ενιαία σκέψη. Ο Φελίπε Γκονζάλες το είπε και τη δεκαετία του 1990 ότι έχουμε μία επιλογή το σωστό πρέπει να το προωθήσουμε και όλα τα υπόλοιπα είναι λάθος και τιμωρούνται. Η επίπτωση είναι ότι εμείς που παίρνουμε τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως ξεχνάει τα προβλήματα που ενέχει και δημιουργεί αυτή η πολιτική. Παραδείγματος χάρη, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Συνένεση έχουν την κοινωνική συνένεση. Όχι, αμφισβητούνται. Η λιτότητα, α πούμε, πλήττει πολύ περισσότερο κάποια κρατημέλη και κάποιε περιφέρειέ του από κάποια άλλα κρατημέλη. Έτσι λαμβάνουμε σήμερα τι αποφάσει μα. Κάποιοι, αν κάποιοι φορεί ε, διατυπώσουν εναλλακτικέ πολιτικέ, τι γίνεται με αυτέ. Διάβασα μία έγγραφα, ε, ένα έγγραφο για τη λιτότητα σε ε, αντιδιαστολή με την ανάπτυξη. Ε, όπου λέει ότι υπάρχει μία συνένεση για έναν, ένα διαφορετικό μοντέλο που δεν θα βασίζεται στη λιτότητα. Ποιος θα το προωθήσει. Θα έπρεπε να ληφθούν οι αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες ε, θα μπορούσαν να είναι ε, διαφορετικές από αυτές που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε το ελληνικό δράμα. Η απόφαση του, οι αποφάσεις του Καραμαλή, όπου ε, δημιουργούνταν προβλήματα για όλους τους πολίτες στην ε, Ευρωζώνη. Τώρα, ε, από τα μοντέλα που υπάρχουν στην Ελλάδα, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα για τους Έλληνες πολίτες. Πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο ταλανίζεται από την ίδια σύγκρουση. Αν δούμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στα εθνικά κοινοβούλια για τους προϋπολογισμούς, τότε λαμβάνονται με βάση το τι θέλουν οι δικοί σας εκλογείς, ο δικός σας λαός. Και οι συνέπειες μπορεί να μην είναι συνεπείς με το σωστό, ε, με βάση τις ε, αξίες και τα θέσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το σύστημα είναι μη βιώσιμο. Και το Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς θέτει αυτό το δίλημα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η λύση λοιπόν. Ίσως η επικουρικότητα. Όμως η επικουρικότητα σημαίνει ότι οι αποφάσεις για τις πολιτικές θα πρέπει να ληφθούν στο πιο αποκεντρωμένο επίπεδο εφόσον μπορούν να προωθηθούν και να τις διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Τι σημαίνει αποτελεσματικά. Χρειαζόμαστε κριτήρια για να αξιολογήσουμε το αποτελεσματικό. Και θεωρώ ότι το κριτήριο είναι ποιος επηρεάζεται από αυτές τις πολιτικές. Ποιος εποφελείται από τα θετικά ή από τα αρνητικά που προκύπτουν από κάποιες δράσεις και κάποιες πολιτικές. Γιατί ορισμένες αποφάσεις επηρεάζουν τον κόσμο πέρα από το κέντρο που λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Μπορούμε εδώ να δούμε τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Αγαθά που έχουν σημασία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτή η θεωρία για τα δημόσια αγαθά μπορεί να μας βοηθήσει ε, για να προχωρήσουμε. Αν επικουρικότητα σημαίνει αποκέντρωση, δηλαδή αποφάσεις ε, λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, είναι πιθανό ότι οι επιρροές ε, αυτών των αποφάσεων στα υπόλοιπα επίπεδα θα αυξηθούν. Αν όμως επικουρικότητα σημαίνει ότι δίδονται αρμοδιότητα σε μια αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων αγαθών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε η επικουρικότητα μπορεί να είναι η απάντηση. Αποτελεσματική διαχείριση σημαίνει καταρχάς μείωση των επιπτώσεων των πολιτικών στα επίπεδα που δεν θέλουμε. Δηλαδή, οι αποφάσει που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο να επηρεάζουν και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ελληνική, α πούμε, κρίση. Οι αποφάσει ε, των Ελλήνων επηρέασαν και του υπόλοιπου, πέρα από του Έλληνε. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε τι αποφάσει για, ε, για τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά που επηρεάζουν κάθε πολίτη. Για να το κάνουμε αυτό, αυτό που χρειάζεται. Και αυτό είναι αντίθετο με αυτή τη φιλοσοφία που σας έφερα εδώ σε αυτό το δωμάτιο, για να ακούσετε αυτή τη συζήτηση είναι η ανάγκη να διαχωρίσουμε τις αρμοδιότητες ανάμεσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο και να μην τις μπλέξουμε, να μην τις ανακατέψουμε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν οι πολίτες, θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές και όχι να ανακατεύουμε τις ευρωπαϊκές με τις εθνικές εκλογές. Το επιχείρημα που θέτω είναι ότι τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά είναι το κριτήριο με βάση το οποίο λαμβάνεται αποφάσεις και με βάση ε, τα οποία επιτρέπεται στον κόσμο να εκφράσει την άποψή του. Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία είναι η απάντηση, δηλαδή ξαναβλέπουμε την, το όλο μας οικοδόμημα. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και μόνο για αυτά και δίνεται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα αποφασίζει και όχι στα κράτη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ζήτω στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας άκουγα πολύ προσεκτικά και ξέχασα να σας διακόψω νωρίτερα. Περνάμε τώρα στον Ντόμινικ Χάνιγκαν, ο οποίος εργάζεται και στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Έχει την ιδιαίτερη ορολογική. Σας δίνω το λόγο αυτής αμέσως. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι προσκεκλημένοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι πραγματική τιμή το, ότι μιλάω σήμερα στην Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το διοργανώνει αυτή την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ήδη είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση το πρωί, η οποία συνεχίζεται και σήμερα το απόγευμα. Το βασικό ζήτημα είναι ποιο πραγματικά μπορεί να καθορίσει το δρόμο για τον άκαμψη τη Ευρώπη. Πώ μπορούμε να αυξήσουμε την ε, δημοκρατική νομιμότητα στα πλαίσια τη οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πώ μπορούμε να επεκτείνουμε την νομιμότητα αυτή, καθώ προχωρούμε σε μια πιο βαθιά ολοκλήρωση. Από ό,τι φαίνεται, όλοι αρχίζουμε και συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα, ενώ ακούγονται πολλέ διαφορετικέ απόψει. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από μόνο το γεγονό ότι οι συζητήσει αυτέ λαμβάνουν χώρα και πραγματικά ελπίζουμε ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να σα πω ότι πρόκειται για το τρίτο φόρουμ στην τελευταία αυτή εβδομάδα, στην οποία είχα τη δυνατότητα να ακούσω τέτοιε συζητήσει και να ανταλλάξω απόψει με του συναδέλφου μου. Συμμετείχα σε ένα άτυπο συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα και επίση ήμουν επικεφαλή τη συνεδρίαση ΚΟΖΑΚ ε, παρουσία του κυρίου Σεφκοβίτς ε, και οι δύο συναντήσεις αυτές στα χώρα στο Δουβλίνο στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας. Κεντρικό ζήτημα και των δύο αυτών συναντήσεων είναι ότι υπάρχει μία ανησυχία όσον αφορά την αύξηση του διακυβερνητικού μοντέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τελικά διαβρώνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική επιτήρηση. Πρέπει να διορθώσουμε το φαινόμενο αυτό. Χρειαζόμαστε ευρωβουλευτέ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος κοινοβουλευτικό έλεγχος. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι εκφράζω αυτή τη στιγμή το δικό μου Εθνικό Κοινοβούλιο, δεν εκπροσωπώ όλα τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είμαι μόνος μου όταν λέω ότι εν γέννη τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν έχουν εμπλεκεί επαρκώς ...στις ε, τελευταίες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη δική μου τη χώρα υπάρχουν κάποιες συνταγματικέ απαιτήσει προκειμένου να γίνονται δημοψηφίσματα για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που εκχωρείται αρμοδιότητα. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και εμείς ένα δημοψήφισμα όσον αφορά την επικύρωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και ξεκίνησε γι' αυτό το λόγο μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ιρλανδία την, τον προηγούμενο χρόνο η δική μου επιτροπή ήταν επικεφαλής της συζήτησης αυτής και είχαμε ομιλητές από όλε τις ε, γωνιές ε, του Ιρλανδικού της Ιρλανδίας και καταφέραμε ουσιαστικά να συλλέξουμε πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το ζήτημα του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Ξέρετε ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο αποτελεί ουσιαστικά μια επανάληψη πραγμάτων που είχαν αποφασιστεί προηγουμένως στην τροποποιημένη από το Six Pack ε, Συμφωνία Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το πρόβλημα όμω είναι ότι τα περισσότερα μέτρα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο ήδη υφίσταντο. Πάρα πολλέ ε, τελευταίε τροποποιήσει στην οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν όμω γίνει κατανοητέ. Και σίγουρα δεν έχουν γίνει κατανοητέ ούτε από πάρα πολλού βουλευτέ εθνικού αλλά και πολύ περισσότερο από του Ευρωπαίου πολίτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τα νέα αυτά στοιχεία που προκύπτουν στην οικονομική διακυβέρνηση να συζητηθούν από τα εθνικά κοινοβούλια. Μόνο στα πλαίσια τη συζήτηση για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία όσον αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο, άρχισε ο κόσμο να συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ποιε είναι οι αλλαγέ. Η όλη αυτή συζήτηση λοιπόν βοήθησε στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η γνώση τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού, ε, Ιρλανδικού λαού όσο και σε επίπεδο Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, η Ιρλανδία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο ζήτημα το οικονομικό. Είναι μία από τις χώρες οι οποίες υποστηρίζεται οικονομικά από τις άλλες χώρες, μία χώρα η οποία προσπαθεί να ανακάμψει και ελπίζει να το πετύχει μέχρι τα τέλη του έτους. Θα το καταφέρουμε να το κάνουμε σε αυτό μόνο αν έχουμε την υποστήριξη των εθνικών βουλευτών και των πολιτών μας και θα μπορέσουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την γνώση μας και να αυξήσουμε και την υποστήριξη αν πραγματικά μπορούμε εμείς ως Ιρλανδικό Κοινοβούλιο να δώσουμε συγκεκριμένε ευθύνε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένω, είμαι σαφώ υπέρ τη συζήτηση αυτή για μια αυθεντική γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα όλα συζητούνται σήμερα, όπω για παράδειγμα το σχέδιο εγγράφου του Νοεμβρίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η, η σχετική έκθεση του κ. Βαν Ρομπέη και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του προηγούμενου μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και ποιε είναι οι ευθύνε των ίδιων των Εθνικών Κοινοβουλίων, πώ μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη πρόταση από τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι κάτι το οποίο μα ανησυχεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα πρέπει επίση να ενισχυθεί ο οικονομικό διάλογο. Πώ μπορεί όμω να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ακούσαμε διάφορε εναλλακτικέ, διάφορε απαντήσει προκειμένου να έχουμε έναν ενισχυμένο διάλογο. Βλέπουμε ότι μια συνεδρίαση σαν τη σημερινή, όπου εθνικοί βουλευτέ έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουν τα ζητήματα αυτά, ένα πολύ θετικό βήμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το όσα είπε ο Επίτροπο Εύκοβιτ στο Δουβλίνο, στη χθεσινή συνεδρίαση τη Κόζακ, ότι θα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επισκέπτεται στο μέλλον πολύ περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα πρόοδου. Χρειαζόμαστε όμω και μια μεγαλύτερη δέσμευση των εθνικών κοινοβουλίων σε πολυμερέ επίπεδο η συνάδελφός μου, η οποία είναι επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην Δανία, διοργάνωσε μια συζήτηση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θέλοντας πραγματικά να ενισχύσει περισσότερο την συμμετοχή των εθνικών βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Από 12 χώρες συμμετείχαν βουλευτές στη συνεδρίαση αυτή. Επίσης, την ε, προηγούμενη εβδομάδα μέλη της δικής μου επιτροπής ε, συνεδρίασαν με ε, Γερμανούς συναδέλφους. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε επαφές ανάμεσα στη δική μου Εθνική Κοινοβουλευτική Επιτροπή με αντίστοιχους συναδέλφους μας από τη Σουηδία. Θεωρώ ότι αυτές οι διασυνοριακές ανταλλαγές, οι ανταλλαγές μεταξύ εθνικών βουλευτών και επαφές μεταξύ αυτών μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στο να καταλάβουμε καλύτερα πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την δημοκρατική επιτήρηση, καθώς επίσης και τη λογοδοσία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης ελπίζω ότι ε, η επόμενη συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοβουλίων που θα γίνει στην Κύπρο πραγματικά θα καταλήξει συγκεκριμένε προτάσει για το πώ μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα ο διακοινοβουλευτικό διάλογο και η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπήρξε ποτέ πιο σημαντικό. Βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλε τροποποιήσει στα πλαίσια τη οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλε αλλαγέ θα έρθουν και στο μέλλον. Ξέρουμε ότι θα έχουμε εξελίξει όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, σύντομα ενδεχομένω να εγκριθεί η νομοθετική δέσμη των δύο μέτρων, το 2 θα πρέπει λοιπόν εμεί, ω εθνικοί βουλευτέ να μας σε θέση να βασιστούμε στη δική μας εμπειρογνωμοσύνη καθώς επίσης και στη γνώση που υπάρχει εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Προκειμένου όμως να κάνουμε κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε την απαραίτητη διάρθρωση, την απαραίτητη αρχιτεκτονική για τη λήψη αποφάσεων. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν επίση και στα πλαίσια τη Προεδρία τη ΚΟΖΑΚ να προωθήσω τα ζητήματα αυτά και στο φόρουμ αυτό. Στη χθεσινή συνεδρίαση τη ΚΟΖΑΚ στο Δουβλίνο αποφασίσαμε ότι στην επόμενη συνεδρίαση τη ΚΟΖΑΚ τον Ιούνιο θα πρέπει να έχουμε μία έκθεση για το πώ εξελίχθηκε η συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοβουλίων στην Κύπρο που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο. Ελπίζω επίση ότι σήμερα το απόγευμα θα ακούσουμε πολύ σημαντικέ συζητήσει και απόψει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Thank um, Ευχαριστώ. Να κάνουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων. Ήδη έχω λάβει διάφορες κάρτες που είναι μόνο από εθνικούς βουλευτές. Παρακαλώ πρέπει να συμπληρώσετε την κάρτα σας στο έντυπο. Δεν πρέπει να σηκώσετε το χέρι σας. Πρέπει να δείξουμε περισσότερη πειθαρχία. Πρώτα λοιπόν Έχουμε τον κύριο Μαρκ Φρανσουά Γάλλο Γερουσιαστή που υπέβαλε πρώτος το αίτημά του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προηγούμενους που τόνισαν ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δημιουργεί ένα χώρο συζητήσεων και υπάρχει ανάγκη αυτού, για αυτόν τον μόνιμο διάλογο μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα πρέπει να δράξουν αυτή την ευκαιρία, τη σημαντική που τους δίνεται τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και νομίζω ότι από πλευράς της Κομισιόν υπήρχε μεγάλη διαθεσιμότητα να έρθουν ενώπιόν μας ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια να λογοδοτήσουν. Ελπίζω αυτή η διαθεσιμότητα να προκαλέσει ανταλλαγές απόψεων χρήσιμες στις χώρες μας. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην ομιλία του κυρίου Κολινιού για το θέμα που αφορά την νομιμοποίηση των πολιτικών μας και το ότι οι εκλογές που λαμβάνουν χώρα στις ε, χώρες μας μοιάζουν με περιορισμένη σημασίας ε, εκλογές που δεν μπορούν να τροποποιήσουν την ενιαία σκέψη που επικρατεί και ότι η Ευρώπη οδεύει προς την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί χωρίς να παίζουν ρόλο οι εθνικές εκλογές. Και τα αποτελέσματά τους δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει πλήρως αυτό. Διότι Ας δούμε τι έγινε τον ε, φθινόπορο του, συγγνώμη, την άνοιξη του 12. Λόγω της νέας αντίληψης ε, που εκφράστηκε για την ανάπτυξη και την αναγκαιότητα πιο δυναμικής αντιμετώπισης του θέματος ανάπτυξης από την εκλογή του Γάλλου Προέδρου Ολάοντα που επιθυμεί η Ευρώπη να ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτές οι εθνικές εκλογές όντως έκανε το δρομέα να αλλάξει θέση. Ίσως με περιορισμένο τρόπο τροποποίησε την ενιαία αυτή αντιμετώπιση του θέματος της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Να λοιπόν πως οι εθνικές εκλογές τροποποιούν τον τρόπο αντιμετώπισης ε, της πραγματικότητας. Άρα δεν είναι ουδέτερες, δεν είναι λίγο χρήσιμες αυτές οι εκλογές. Ακόμη και αν μπορεί να αλλάξει η ενιαία αντιμετώπιση, είναι σαφές, όπως είπαν ορισμένοι, ότι ο τρόπος αντίδρασης τη Ένωση πρέπει να βελτιωθεί. Γιατί οι καταστάσεις αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει λοιπόν να αντιδρούμε πολύ γρήγορα. Το βλέπουμε και για το θέμα των ρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και για τα δημοσιονομικά θέματα της Ευρώπης. Οπότε πώς αυτή η ταχεία αντίδραση θα έχει την αναγκαία αποδοχή. Πώς οι ενέργειες που αναλαμβάνουμε θα έχουν την αναγκαία δημοκρατική νομιμοποίηση και αποδοχή λόγω και της περιπλοκότητας των θεμάτων, όπως υπόθηκε, που περιορίζουν τις επιλογές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξηθεί ο έλεγχος από τα Εθνικά Κοινοβούλια Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η διαφορά φάση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρώπη που ήδη έχει καταγγελθεί θα αυξηθεί περαιτέρω. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε την ε, διάθεσή της. Εμείς ως Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίδεται. Ανά χώρα λοιπόν να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και δημοκρατική επικύρωση των αποφάσεων που λαμβάνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο επόμενος από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Γιώχιμ Σπέτς, που είναι στην Επιτροπή για τις ε, Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, να απαντήσω στον κύριο Βόλφ, που είπε «Ζήτω Ευρωπαϊκή Δημοκρατία». Βίβλα, και Ευρωπαίν. Συμφωνώ αλλά δεν ξέρω πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα δέχονταν αυτό του το σύνθημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν θα επιτύχουμε ουσιώδη μεταφορά κυριαρχία στον τομέα της οικονομικής πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής προς την Ένωση. Το επόμενο βήμα πιστεύω πρέπει να είναι η Ευρώπη να εγγυηθεί μία αξιόπιστη συνεργασία των κρατών μελών με την επιτήρηση της Κομισιόν, ούτως ώστε να τηρούνται οι αμοιβαίως ε, δοθήσεις υποσχέσεις, όχι όπως δηλαδή με τη συνθήκη του Μάστριχτ, διότι αλλιώς θα χαθεί η εμπιστοσύνη, που είναι βάση για οποιαδήποτε μεταφορά κυριαρχίας. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ως πίεσης από τους ομοτήμους, θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε μία αξιόπιστη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Βεβαίως υπάρχει σύγκρουση διαφορετικών λογικών, αλλά δεν έχουμε καμία δυνατότητα, τουλάχιστον ενδιαμέσως, παρά να έχουμε μία κυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Μια διακυβέρνηση σε πολλαπλά επίπεδα. Διότι βεβαίω, βεβαίω, έχει γίνει η συζήτηση. Θέλαμε την κοινοτική μέθοδο στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο εμείς στη Γερμανία. Αλλά δύο κράτη-μέλη το απέρριψαν οριστικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Η απάντησή μας ήταν το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι ενδιάμεση συμβατικά λύση με προοπτική φυσικά κάποια στιγμή να περάσουμε στην κοινοτική μέθοδο. Ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα. Ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Εξακολουθούν να εφίστανται εθνικές κοινέ γνώμες. Ο πολιτικός διάλογος στις χώρες μας γίνεται σε επίπεδο κράτους. Και όποιος έχει συμμετάσχει έστω και μία φορά στις ευρωεκλογέ, ξέρει ότι και οι ευρωεκλογέ καθορίζονται και κυριαρχούνται από εθνικά και όχι ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό είναι λυπηρό, πρέπει να προσπαθήσουμε να το τροποποιήσουμε, αλλά πρέπει προς το παρόν να εργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο. Βεβαίως μου αρέσει ε, η νέα αυτή αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, πολυμερείς σχέσεις συμβατικές υπό την επιτήρηση της της Κομισιόν με την καλύτερη κοινοβουλευτική επιτήρηση. Βεβαίω είναι του mixtum μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων αυτό που έχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με τους ομιλητές. Θα ακούσουμε και έναν τρίτο εθνικό βουλευτή αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γαλλικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Καρές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές που παρουσίασαν με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τις απόψεις τους, με τρόπο που εγείρει ερωτηματικά. Η κατάσταση είναι νέα Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα. Αλλάζει η εποχή μας, αλλάζουν τα δεδομένα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η συνθήκη, η δημοσιονομική συνθήκη και το πακέτο των δύο μέτρων, το 2 πακ, δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούμε για, τα, για τις προτινόμενες αλλαγές και αυτές που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλλαγή είναι πολύ σημαντική. Έχω την εντύπωση ότι στα πλαίσια αυτής της κρίσης έγινε μια μεταφορά κυριαρχίας, την οποία δεν έχουμε χωνέψει σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά έχει γίνει όμως. Τα εθνικά κοινοβούλια, οι εθνικοί βουλευτές, ως συνέπεια, πρέπει να εφαρμόσουν κάποιες αποφάσεις ή κάποιους προσανατολισμούς που ελήφθησαν αλλού, σε άλλο κέντρο λήψη αποφάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι απλώς δημοσιονομικές αποφάσεις. Όταν ε, κοιτάμε τα κείμενα της Κομισιόν, η ετήσια εξέταση για την ανάπτυξη ή οι προσανατολισμοί που είναι συστάσεις που προτείνει η Κομισιόν για κάθε χώρα. Όλα αυτά τα έγγραφα καλύπτουν το σύνολο της οικονομικής πολιτικής και της κοινωνικής πολιτικής. Ακόμα και τα συνταξιωτικά συστήματα ε, τίθενται ένα αμφιβόλο. Ο εργασιακός κώδικας. Μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων και όχι μόνο ε, για κάποιους δημοσιονομικούς δείκτες. Γίνεται μια ριζική λοιπόν αλλαγή και είμαστε ενώπιόν της. Θα πρέπει λοιπόν να διερωτηθούμε για το θέμα της δημοκρατίας. Υπάρχουν δύο θεσμικά όργανα σε αυτό το σύστημα που αποφασίζουν τελικά και που δεν λογοδοτούν στην πραγματικότητα. Είναι η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Η Κομισιόν δεν λογοδοτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάποια θέματα, ιδίω για τα δημοσιονομικά, και το Συμβούλιο, σίγουρα οι χώρε, ή μάλλον οι κυβερνήσει λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών του κοινοβουλίων, αλλά όταν συνέρχεται το Συμβούλιο, συναποφασίζουν εκεί οι χώρε. Και αν μια χώρα θέλει να διαφύγει από αυτό το πλαίσιο πειθαρχία, δεν μπορεί πλέον να το κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αυτό το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας. Άκουσε αυτό που είπε ο κύριος Βόλφ. Τον τρίτο άξονα δεν τον ανέπτυξε επαρκώς. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να επιτρέψουμε τη μετεξέλιξη των θεσμικών μας οργάνων. Και ελπίζω ο κύριος Βόλφ να μου απαντήσει. Σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα, τα ομοσπονδιακά θεσμικά όργανα ελέγχουν Έχουμε ένα σύστημα όπου τα, θεσμι... ομοσπονδιακά θεσμικά όργανα ελέγχουν τα τοπικά θεσμικά όργανα. Στην Αμερική, ας πούμε, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Καλιφόρνιας. Εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα λοιπόν εμείς. Ίσως θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά θεσμικά όργανα, όχι αμυγός ε, ομοσπονδιακά. Ίσως μέσω της ε, πλήρους Συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι αυτό τον άξονα θα πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω. Η Άννη από τους Σοσιαλιστές, Ευρωβουλευτής. Θα μιλήσω ε, ελληνικά. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ε, αυτή η συζήτηση. Θέλω να επισημάνω ε, ότι είμαι Ελληνίδα Ευρωβουλευτής. Είμαι λοιπόν ένα ζωντανό παράδειγμα του ελληνικού δράματος που είπε και ο κύριος ε, ε, Κολινιό. Ε, κύριε Γουλφ, είπατε στην τοποθέτησή σας και πολύ σωστά ότι η διαδικασία λήψης των αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης προσδιορίστηκε και προσδιορίζεται από τις πιέσεις των αγορών και από τα όρια που θέτουν οι συνθήκες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εξ αντικειμένου αυτό σημαίνει ότι είχαμε μια κατάσταση όπου είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στην ταχύτητα και την δημοκρατία. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και ε, όχι μόνο, είχαμε να διαλέξουμε επίσης ανάμεσα στην αποδοχή και εφαρμογή των αποφάσεων ή τη χρεοκοπία. Άρα, ε, εκτός από τα externalities, κύριε Κολυνιό, που είχαν ασφαλώς και αδιαμφισβήτητα οι αποφάσεις για την Ελλάδα, υπήρχαν και πολύ σοβαρά internalities, διότι στην ουσία και στο εθνικό επίπεδο, σε πολλά κράτη-μέλη, αυτά που ήταν κυρίως στο επίκεντρο της κρίσης, ε, η διαδικασία της δημοκρατικής λογοδοσίας και του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων είχε εντελώς εξαφανιστεί. Αυτό με την σειρά του συνδέεται με την κοινωνική αποδοχή των πολιτικών και των προγραμμάτων. Η κοινωνική αποδοχή μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται όλο και πιο ε, μικρή και τελικά υπονομεύεται η ίδια η υλοποίηση των συμφωνημένων πολιτικών και είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Θέλω λοιπόν να κάνω δύο ερωτήματα. Άκουσα τις προτάσεις σας. Ε, ασφαλώς το ευρωπαϊκό εξάμεινο μπορεί να συμβάλλει αλλά μήπως τελικά μιλάμε για ημίμετρα μέχρι να φτάσουμε κύριε Κολυνιό στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος προφανώς να το λύσουμε αυτό το ζήτημα με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Και τελικά τα σημερινά μας κοινοβουλευτικά μοντέλα, οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες στην Ευρώπη σήμερα είναι συμβατές με την παγκοσμιοποίηση ή πρέπει να ξαναδούμε στην ουσία από την αρχή τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στα κοινοβουλευτικά μας συστήματα που είναι βασισμένα στο κράτος έθνος και το κράτος έθνος ε, με σαφήνεια ε, σε εποχές παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να ανταποκριθεί οι δομές τους στις προκλήσεις που έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you and από τη Λιθουανία, ο κύριος Ζεματάτης. E, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Ή μάλλον θα ήθελα να μιλήσω λίγο αργότερα, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ήταν αυτή η σειρά με την οποία ζητήσατε να μιλήσετε. Εντάξει, αν το κάνω αυτό για όλους θα υπάρξει πρόβλημα. Από η Μέρι Βαντελίντεν από την Ολλανδική Γερουσία είναι η επόμενη. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω το λόγο στον προηγούμενο μιλητή λίγο αργότερα. Ευχαριστώ. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι ότι δεν συμφωνούμε όλοι για το είδος της Ευρώπης που θέλουμε. Υπάρχουν χώρες που θέλουν μια Ευρώπη ελευθέρων συναλλαγών και μια ε, Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα επιλέγουμε ό,τι θέλουμε από το μενού. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ένα μενού με 27 πιάτα, με 27 ορντεύρ, με 27 γλυκά. Θα πρέπει να επιλέξουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να καταδείξει στον κόσμο τα επιτεύγματά της. Μέχρι στιγμή δεν το έχουμε κάνει και δεν μπορούμε να το κάνουμε όσο είμαστε διαιρεμένοι. Όταν οι διαδικασίες λήψη των αποφάσεων είναι αδιαφανεί. θα ήθελα να κάνω έκκληση λοιπόν για να ενισχύσουμε το Eurogroup, το Eurogroup. Είναι ένας ε, μοχλός ενσωμάτωσης, ολοκλήρωσης. Είναι ε, ένα μέσο ολοκλήρωσης ακόμα και, τις, ε, και για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Ανήκουμε σε ένα κλαμπ. Όταν ανήκουμε, ας πούμε, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δεχόμαστε τους κανόνες του παιχνιδιού. Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε ακολουθώντα κάποιου κανόνε. Ακόμα και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να του μάθουν αυτού του κανόνε. Δυστυχώ, αυτά τα εθνικά κοινοβούλια ε, εμπλέκονται όλο και περισσότερο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν. Όταν είμαστε μειονότητα, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με κάποια πράγματα, θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε. Γι' αυτό νομίζω ότι το σχέδιο Φανρόμπουι είναι ένα θαυμάσιο πρόγραμμα για το μέλλον. Και αν χρειάζεται με περισσότερη... Και αν υπήρχε στην Ευρώπη μεγαλύτερη πεποίθηση για όλα αυτά τα πράγματα, μεγαλύτερη συνένεση, θα προχωρούσαμε πιο απρόσκοπτα. Είναι δύσκολο να πείσουμε τον πολίτη ότι του ετοιμάζουμε ένα ροζ μέλλον με αυτόν τον τρόπο. Μιλήσατε για την εθνική κυριαρχία. Σίγουρα είναι πιο περιορισμένη η κυριαρχία των κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει οι μεν να πάρουν στα σοβαρά τους δε. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν και εμπιστοσύνη τα εθνικά κοινοβούλια. Και όταν οι εθνικοί βουλευτές έχουν εμπιστοσύνη, τότε προωθούν και το ευρωπαϊκό, τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την ευρωπαϊκή άποψη. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ολλανδία. Έχουμε την Άνω και την Κάτω Βουλή. Έχουμε τη Γερουσία και έχουμε και τη Βουλή. Και η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία όσο δεν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα της Βουλής. Εγώ εδώ και χρόνια είμαι, ήμουν υπέρ της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ασκώντας όμως κάποιες επικρίσεις. Και πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ανοιχτό στις κριτικές, ακόμα και αν η κριτική στρέφεται εναντίον του. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στη Βουλή των Λόρδων. Πάρισον. Κυρία Πρόεδρε, για 14 χρόνια συμμετέχω στην Επιτροπή στο, του Εθνικού μου Κοινοβουλίου. Συμμετείχα όμως επίσης και σε αυτό το κοινοβούλιο και θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε την ακρόαση, ότι είχαμε μια ακρόαση καθώς επί για τον Αλεξάνδρ Λαμφαλουσί, θυμάμαι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θυμάμαι την ημέρα που κάναμε την ακρόαση για την επιλογή του και θυμάμαι τότε ότι είχα εκδώσει και ένα δελτίο τύπου λέγοντας ότι ε, η Ευρώπη επέλεξε τον νέο τραπεζικό της διευθυντή διαχειριστή και κανείς τότε δεν έδειξε καμία απολύτως σημασία. Έκτοτε όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει ακόμα και οι ευθύνες και αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εμεί ως εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει πλέον να προετοιμαστούμε για τις μελλοντικέ προκλήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα από την εκπρόσωπο της Bundestag το γεγονός ότι πήγε ο Μάριο Ντράγκη εκεί και, και εμείς ε, όταν ε, εκδώσαμε την έκθεσή μας για την Τραπεζική Ένωση, είχαμε κάνει μία τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βοηθός του Μάριου Ντράγκη. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε μια επαφή ανάμεσα στους εθνικούς βουλευτές και εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που παίρνουν πολύ σημαντικές αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα στην ε, Βουλή των Λόρδων κάνουμε και ένα σεμινάριο για την πολιτική δημοσιονομική λιτότητα, όπου εκεί πέρα συζητάμε πώ μπορούμε να ανταποκριθούμε στι νέε οικονομικέ συνθήκε. Πρέπει να σα πω ότι αποφασίζοντα το νέο πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουμε, ο επικεφαλής της ε, Αρμόδιας επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη Βουλή των Λόρδων απευθύνθηκε σε εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων προσπαθώντας να αποφασίσει τελικά τι πρέπει να κάνουν τα κοινοβούλια και πώς πρέπει να συμμετέχουν. Και πιστεύουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει πραγματικά να βρίσκονται σε μια γνήσια επαφή μεταξύ τους, να κάνουν μια γνήσια ανταλλαγή απόψεων, να χρησιμοποιήσουν ακόμα και τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Βόλφ, αν μπορεί να μας πει λίγα περισσότερα πράγματα για το τι μπορεί να γίνει για την Ευρωζώνη, πώς μπορούμε να έχουμε εμεί ένα πιο αποτελεσματικό έλεγχο και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τελικά ο έλεγχος αυτός να γίνεται μόνο από κράτη-μέλη που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι μια σχετική απόφαση λήφθη στις 18 Δεκεμβρίου. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τον Ντομινίν Χάνιγκαν να μας μιλήσει λίγο περισσότερο για τη σημασία που θα γίνει από τις 21 μέχρι τις 22 Απριλίου, δηλαδή τη διάσκεψη των Προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων τι είδους προτάσεις θα πρέπει να γίνουν βάσει των σημερινών συζητήσεων, έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν πραγματικά και επιτυχώς στην όλη αυτή διαδικασία την οποία θέλει να προωθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μπορούμε δηλαδή ως εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουμε πραγματικά αυτά τα οποία αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι στις 18 ε, Δεκεμβρίου το Συμβούλιο προχώρησε κάποιες αποφάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο τριμερούς διαλόγου. Πρέπει λοιπόν να δώσει και το Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη του, ιδίω όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή επιτήρηση των Τραπεζών. Δεν έχει ληφθεί κάποια επίσημη απόφαση. Πρέπει να σα πω ότι με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η απόφαση αυτή, η αρχική πρόταση θα τροποποιηθεί, ελπίζουμε, ικανοποιητικά. Περνάμε τώρα στην Φιλανδία, στον επικεφαλής ε, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ο κύριος Κοσκάνεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πάρα πολλές απόψεις όσον αφορά την εθνική κυριαρχία, όσον αφορά το νέο αυτό πλαίσιο το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει πραγματικά να δυναμώσει την θέση της στο παγκόσμιο αυτό προσκήνιο. Πρέπει πραγματικά να καταφέρουμε στα πλαίσια του νέου αυτού πλαισίου το οποίο προκύπτει να διασώσουμε και εμείς την εθνική μας κυριαρχία και να καταφέρουμε επίσης να ενισχύσουμε κάποιες αρμοδιότητες των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπουμε πολύ συχνά ότι η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε μια συρρήκνωση της ε, συλλογικής κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είδαμε ότι ε, σε ορισμένε περιπτώσεις ε, η συλλογική μας κυριαρχία μπορεί πραγματικά να αυξηθεί, αρκεί όμως να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις και πρέπει αυτόν να το συνειδητοποιήσουμε σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Όσον αφορά τώρα τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και εξουσιών, θα πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ξέρετε ότι γίνονται συστάσεις αναχώρα και θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις γενικές οικονομικές κατευθύνσεις που δίδονται προς τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχουν αποκλήσεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Οι απόψεις αυτές επηρεάζονται πολλές φορές και από το πολιτικό φάσμα, αλλά υποστηρίζει δεξιά, αλλά η αριστερά. Πιστεύω πάντως ότι οι συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνονται, πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απαραίτητα πάντα αντικειμενική. Καταλαβαίνετε ότι πολλέ φορέ κρύβεται και πίσω από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμα μια κάποια πολιτική άποψη. Θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εντείνει τον διάλογο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω όταν αυτή εκδίδει ειδικέ αναχώρα τάσει. Επίση, πιστεύω ότι στα πλαίσια τη δική μα συνεδρίαση τώρα θα πρέπει να δούμε βάσει ποια γνώση και εμπειρογνωμοσύνη τελικά μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει συστάσει για τα κράτη-μέλη. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια των συστάσεων αυτών να βγόταν και η φωνή των εθνικών κοινοβουλίων. Και θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζει τελικά τι πιστεύουν, τι πρεσβεύουν οι εθνικοί βουλευτέ. Και θα πρέπει να ακουστούν βέβαια και οι απόψει δεξιά πάλι, αλλά και οι απόψει τη αριστερά προκειμένου να καταλάβουμε τελικά ότι ε, δίστανται οι απόψεις, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την νομοθεσία που έχει να κάνει με την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτή λοιπόν την ε, ανταλλαγή απόψεων και σε αυτό το μηχανισμό που θέλουμε να εγκρίνουμε για την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο, πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες επαφής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, τις ήδη καλές γνώσεις που έχουμε ως Εθνικά Κοινοβούλια να τις αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Εν κατακλείδη, όσον αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ως προς αυτό τι είναι το πιο σημαντικό. Ο δημοκρατικός έλεγχος βέβαια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μια σχετική μνήμα έγινε όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση πριν από λίγο από ένα συνάδελφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε εμεί να εξασφαλίσουμε αυτόν τον έλεγχο. Οι εξουσίε όμω όσον αφορά την οικονομική και νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν αυξηθεί εξαιτία τη κρίση. Γι' αυτό ακριβώ όμω το λόγο χρειαζόμαστε και εμεί τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταφέρουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε τον πολιτικό έλεγχο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μεγαλύτερη λοιπόν συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον τομέα αυτό. Ξέρετε ότι για παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της διαβούλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικός αυτός έλεγχος. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρι Σμιτ. Ευχαριστώ. Είμαι φιλελεύθερος από τη Σουηδία. Στον Ολλανδό συνάδελφο θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ της ε, ένταξης της Σουηδίας ε, στο ευρώ, αλλά χρειάζομαι την υποστήριξη της πλειονότητας των συμπολιτών και πολλές φορές αισθάνομαι περισσότερο μοναξιά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό που ακούσαμε από τους ομιλητές. Ε, κύριε καθηγητά Κολίνιο, είπατε ε, δημοκρατία της Ευρώπης ή, Γαλλική, ή Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Η καγκελάριος Μέρκελ είχε έρθει εδώ τον Νοέμβριο πηγαίνοντας να συναντήσει τον κύριο Κάμερον και μας είπε ότι ίσως η ευρωπαϊκή ενοποίηση να πρέπει να γίνει βήμα το βήμα να μην ε, απομακρυνθούμε υπερβολικά από τους πολίτες. Έχει επιδείξει ιδιαίτερη επιδεξιότητα και σύνεση θα έλεγα. Αυτό πρέπει να κάνουμε που προτείνει. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ομφαλός της γης εμείς εδώ. Φυσικά, λογικό να το θεωρούμε. Αλλά ακόμη και οι εθνικοί βουλευτές όπως εσείς ε, πρέπει να βοηθήσετε γιατί έχετε βασική αρμοδιότητα. Έχω υπάρξει και εγώ εθνικός βουλευτής. Εμείς είμαστε πολύ πιο κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό πιστεύω, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την εμπειρία μου, πρέπει να μας εμπλέξετε και εμάς στις προσπάθειες. Γιατί ο καθένας κατηγορεί τον άλλον. Στα Εθνικά Κοινοβούλια λένε οι Βρυξέλλες ε, τα κάνουν όλα μουσκεμα. Και κάποιοι εξημών μπορεί και να λένε ότι για 20 χώρες υπάρχει ενδεχόμενο διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ίσως κάποιοι από εμάς να φταίνε γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν να τα πετύχουμε όλα μόνοι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σπέτς. Με συγχωρείτε που μιλάω άσχημα αγγλικά. Είναι άσχημο αυτό. Γιατί το θέμα είναι γενικότερα το θέμα της γλώσσας. Θέλω να κάνω έκκληση σε εσά. Δεν ξέρω εάν συμβαίνει παντού στην Ευρώπη αυτό που προτείνω, αλλά στη χώρα μου δεν συμβαίνει. Επιτρέψτε στην εθνική κοινή γνώμη να μας ακούσει και μας. Αφήστε μας να μιλήσουμε. Φυσικά και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό είναι καλό, αποτελεσματικό. Αλλά θα μπορούσαμε να συναντηθούμε και στα εθνικά σα κοινοβούλια, να έρθουμε ορισμένοι από εσά να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ούτω ώστε να μπορέσουμε, μιλώντα τη γλώσσα μα ο καθένα στις πρωτεύουσέ μας, να κάνουμε πιο ουσιαίο διάλογο. Παρακαλώ ανοίχτε μα την πόρτα. Πρόεδρο. ευχαριστώ. Ίσως τώρα ο κύριος Ζεμετάτης ε, θα ήθελα να συμμετάσχει τώρα από τη Λιθουανία. Α, έφυγε. Α. Α. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, σήμερα θίξαμε μια σειρά από ζητήματα ιδιαίτερα επίκαιρα. Επίκαιρα και για τα εθνικά μας κοινοβούλια και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που μας καλέσατε σε αυτήν την συνάντηση και που μας δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για την Ευρώπη και για το πώς πρέπει να την αλλάξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στην ε, παρουσίαση της κυρίας Φερέιρα που ε, θίγει μια σειρά θέματα που μας ενδιαφέρουν στην ε, προσπάθειά μας για μια πιο ενοποιημένη Ευρώπη, πιο κοντά στους λαούς της. Εάν θέλετε οι λαοί μας να ξέρουν περισσότερα για την Ευρώπη, τότε πρέπει να βοηθήσουν διαδίδοντας τη γνώση για την Ευρώπη τα εθνικά κοινοβούλια, για παράδειγμα, για τα κοινωνικά ωφέλη από την ε, λειτουργία της Ευρώπης. Βεβαίως, κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αλλά το θέμα που ουσιαστικά τίθεται είναι τι ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε απασχόληση ή θέλουμε ένα τεράστιο ε, αριθμό εργαζομένων που ουσιαστικά ε, δεν συμβάλλουν στην οικονομία. Για τα μεγάλα ε, έργα υποδομών. Αποφασίσαμε, είναι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το εάν θα χτίσουμε καινούργια πυρηνικά εργοστάσια ή για εάν θα διακόψουμε τη λειτουργία τους αλλά δεν τους εξηγούμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τι ακριβώς αποτέλεσμα θα έχει η δημιουργία ή η πάυση λειτουργίας ενός πυρηνικού εργοστασίου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα σχετίζεται με τις ευρείες συζητήσεις που κάνουμε για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Αλλά δεν προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να επιτύχουμε την αύξηση αυτής της αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό είναι χρήσιμες οι συζητήσεις όπως οι σημερινές. Καταλήγοντας, θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους να επιτύχουμε περισσότερο, περισσότερη διαφάνεια, ευρύτερο διάλογο μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, θεσμών της Ένωσης γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θέλουν και άλλο το λόγο. Μου μένουν δύο μιλητέ. Γιώργεν Κλούιτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά Μπέρναρντ Ντουκέν από την Ιρλανδία και ίσως και εγώ. Πρώτος λοιπόν ο Γιούργεν. Ευχαριστώ Σάρων. Δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, ο Ολλανδός συνάδελφος είπε ότι πρέπει να βελτιώσει κάπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πολιτική δαπανών, τους, δαπανών του και ότι έπρεπε να υπάρχει περισσότερη κριτική γι' αυτό. Γίνεται κριτική γι' αυτό. Αλλά ποιε είναι οι συγκεκριμένε επικρίσει, θα ήθελα να μάθω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτον, έχει σχετικά περιορισμένο προπολογισμό και είναι μόνο 6% των δαπανών οι διοικητικέ δαπάνε. Για όλα τα κοινοτικά όργανα, για τα κτίρια, του μισθού, τα υπόλοιπα είναι χρηματοδοτήσει που δίδονται στι ε, χώρε μέλη. Αν θέλουμε λοιπόν να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε ανοιχτά. Αλλά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ποια είναι η επίκριση. Πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Και δεύτερον, έχουμε τον τριμερή διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής. Και συχνά ακούμε σε αυτές τις συζητήσεις το Συμβούλιο έχει πολύ πιο περιορισμένες φιλοδοξίες από, τους, ε, από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο προχωρημένο, πολύ πιο κοντά στις απαιτήσεις των πολιτών, αλλά στις εσωτερικές διαπραγματεύσεις το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, συγγνώμη, που φυσικά έχει πολύ πιο ισχυρό ρόλο, περιορίζει την αποτελεσματικότητα των ε, ενεργειών του Κοινοβουλίου. Δεν κάνει αρκετά το Συμβούλιο προς το συμφέρον των πολιτών. Θα έπρεπε λοιπόν ακριβώς τα Εθνικά Κοινοβούλια που συμφωνούν με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επηρεάζουν περισσότερο τις κυβερνήσεις. Μόνο έτσι θα μπορούσε να προχωρήσει συνεργασία. Θα ήταν κάτι τέτοιο χρήσιμο. Αναγκαίο θα έλεγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να συγχαρώ τον Ντόμινι Χάνεκαν για την παρουσίασή του. Ε, παρουσίασε την Ιρλανδική Σκοπιά και δείχνει πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση μια μικρή χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι, που θέσατε είναι ποιος θέτει την πορεία εδώ. Είναι τα Εθνικά Κοινοβούλια, η Κομισιόν, το Συμβούλιο. Η απάντηση είναι απλή. Όλοι μαζί. Σε συνεργασία και διαβούλευση ημέν με τους δε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ είναι ότι γίνεται διαβούλευση, γίνεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πολύ σπάνια έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε αυτό το επίπεδο. Ε, ανταλλάσσουμε απόψεις με τους Υπουργούς, με το Συμβούλιο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πολύ σπάνια συνομιλούμε μεταξύ μας. Ο κύριος Πέτς, ο Γερμανός συνάδελφος, είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τα οικονομικά θέματα. Κάποιος πρέπει να μου πει τι εναλλακτικέ υπάρχουν για χώρες όπως η Ιρλανδία. Είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ της λιτότητας και κάτι άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποιες ήταν οι εναλλακτικέ μας λύσεις. Μα είπαν με έμφαση αυτό έπρεπε να κάνουμε και έπρεπε εμεί να ανασκουμποθούμε και να το κάνουμε. Και το κάνουμε με κόστος και τίμημα και συνεχίζουμε να το κάνουμε κόστο και τίμημα. Είναι σημαντικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια και όλοι οι συνάδελφοι στα άλλα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν τις θυσίες που κάνουμε για το κοινό καλό, για το μέλλον της Ευρώπης, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο για τους Ιρλανδούς. Θα πρέπει λοιπόν τα θεσμικά όργανα να έρθουν στα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να έρθουν πιο κοντά στο λαό μας και να μας εξηγήσουν γιατί να μας εξηγήσουν ποιες είναι οι πολιτικές συνέπειες αν δεν εφαρμόσουμε αυτά που μας επιβάλλονται. Πάνω από 30 χρόνια θέλω να σας πω ότι ήμουν ε, Ιρλανδός βουλευτής και είδα καλά και κακά πράγματα. Και Έμαθα πολλά. Ένα από αυτά που έμαθα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε μαζί με ομοφωνία για το κοινό καλό, να αναγνωρίσουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες ο ένας του άλλου προς το κοινό στόχο με βάση κάποια κοινά πράγματα που όλοι μαζί θα συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Σε λίγο θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μας οι οποίοι θα απαντήσουν στις πολλαπλές αυτές ερωτήσεις που ακούστηκαν. Θα ήθελα όμως πριν να πω ότι όταν ετοιμάσαμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Six Pack, όλα αυτά τα πολύ επιτακτικά ε, νομοθετήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε σε αδιέξοδο. Κάτι που συνέβη και στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, ειδικά για τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου οι γραφειοκράτες τελικά αποφασίζουν τις ε, τροποποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις. υπάρχουν διάφορα θέματα, τα θέματα της ρευστότητα, το CRD και τα λοιπά, που σπάνια συζητιώνται, σπάνια έρχονται οι υπουργοί να συζητήσουν. Δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία, επαρκής έλεγχος. Ε, εξού και οι διαφωνίες. Ε, για τα τραπεζικά ομόλογα, ας πούμε, υπάρχουν διαφωνίες. Ε, και γιατί υπάρχουν διαφωνίες, γιατί δεν ξέρουμε επαρκώς τα δεδομένα. Και ακούγονται διάφορες ιδέες, κυκλοφορούν διάφορες ιδέες. Συχνά εγώ χρειάστηκα να δώσω εξηγήσει σε διάφορες επιτροπές Αυτό θέλω να το τονίσω. Είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι συζητήσει. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρθει σε περισσότερη επαφή με τα κράτη-μέλη για όλα τα νομοθετήματα. Έχουμε ακόμα 25 λεφτά στη διάθεσή μας. Θα, δώσω το λόγο σε άλλους δύο βουλευτές. Ή μάλλον όχι. Άλλαξα γνώμη. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές μας για πέντε λεφτά στον καθένα για να απαντήσουν στα πιο σημαντικά ερωτήματα. Και εν συνεχεία θα ακούσουμε τις καταληκτικές ε, παρατηρήσεις από τους υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές. Να απαντήσετε με την ίδια σειρά με την οποία μιλήσατε, ο κύριος Βόλφ. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω στα γερμανικά στους γερμανούς συναδέλφους. Κύριε Σπάτς, η ερώτησή σας αφορά περισσότερο τον κύριο Κολίνιο, όχι εμένα. Ε, δεν είπα εγώ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ωραία. Παρ' όλα αυτά όμως, θα ήθελα να δράσω συντόμως από αυτού. Νομίζω ότι μια σταδιακή προσέγγιση από πολλές απόψεις είναι καλύτερη. Διότι εσείς είστε πολιτικοί, εσείς μπορείτε να εκτιμήσετε σε τι βαθμό οι πολίτες ε, συμφωνούν μαζί σας, μπορούν να δεχθούν αυτά που προτείνετε. Βεβαίως, δεν μίλησα κατά του, της ΟΝΕ και του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Είναι βήματα αυτά. Αλλά τόνισα ότι είναι ενδιάμεσα βήματα. Να μην έχουμε την αυταπάτη ότι είναι η τελική κατάσταση. Και τονίζω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι μια επιβραδυμένη διαδικασία τόσο μεγαλύτερο κόστος θα έχει. Όσο αργότερα πηγαίνουμε τόσο αυξάνονται από πλευράς του κόστους για το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να τα υποτιμούμε, να μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες. Ότι δεν υπάρχει πια πίεση των αγορών, μπορούμε να χαλαρώσουμε. Τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Θα έκανα λοιπόν έκκληση και περαιτέρω να είμαστε σε στενή επαφή με τους πολίτες για να τους πείσουμε ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα. Τώρα απαντώντας ε, στον, στην Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, το θέμα της κοινωνικής αποδοχής είναι βέβαια πολύ σημαντικό, αλλά πέρα από αυτό, και εδώ να μην έχουμε αυταπάτες ακόμη και αν έχαμε μια πλήρως ομοσπονδιακή ευρωπαϊκή δημοκρατία όπως ε, το έθεσε ο Στεφάν θα έπρεπε να γίνουν επίσης αρκετές προσαρμογές ε, οδυνηρές για την Ελλάδα. Εάν λοιπόν είχε υπάρξει μια τεράστια κρίση στην πολιτεία της Πενσιλβένια, αν είχε καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα και η χαλιβουργία, φυσικά ο λαός της Πενσιλβένια θα είχε υποφέρει πολύ. Η διαφορά όμως είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Πενσιλβένια σταθεροποιείται μέσω του συστήματος των ΗΠΑ και είναι πολύ πιο ευέλικτη η αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι πηγαίνουν σε άλλες πολιτείες. Μην γελιόμαστε λοιπόν. Τα βήματα που πήραμε υπέρ αύξησης ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικά και για ένα κοινό αλλά το θέμα είναι πώς θα μάθουν να ζουν οι πολίτες σε αυτή την ένωση. Θα υπάρχουν περισσότερα μεταναστευτικά ρεύματα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πανάκια βέβαια, αλλά οπωσδήποτε θα ήταν μικρότερες επιπτώσεις ε, της κρίσης. Αλλά βεβαίως η κοινωνική αποδοχή είναι το πραγματικό πρόβλημα και με φοβίζει η κατάσταση όταν ε, βλέπω τι ποσοστά ανεργίας έχουμε στην Νότια Ευρώπη μπορεί να πυροδοτήσουν περαιτέρω προβλήματα. Θέλω να απαντήσω προς τους Γάλλους ε, βουλευτές, άμα επιτρέπετε στα γαλλικά. Το θέμα της κυριαρχίας ε, το υποτιμάτε στη Γαλλία, νομίζω. Αυτή τη στιγμή εντάσσεται κάποιο σε μια νομισματική ένωση, χάνει την ανεξαρτησία του για την νομισματική πολιτική. Αλλά και εν μέρη χάνει την ανεξαρτησία του για την δημοσιονομική πολιτική. Ο πρόεδρος Ολάντ δεν έχει την ελευθερία να διαμορφώσει τον προϋπολογισμό όπως θέλει. Κάνει μια προσαρμογή πολύ σημαντική, προφανώς. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει και την κυριαρχία της Γαλλίας. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν επί του θέματος αυτού και αν θέλουμε να περάσουμε σε μεγαλύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση που τελικά είναι κάτι το απαραίτητο για να συμπληρώσουμε την νομισματική ένωση θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εγκαταλείπουμε ένα τμήμα της κυριαρχίας μας, της εθνικής μας κυριαρχίας. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα είναι το θέμα της κοινοτικής μεθόδου, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία θα πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να περάσουμε στη δημοσιονομική ολοκλήρωση. Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Δεν μίλησα πολύ για, την, για το ομοσπονδιακό όρομα, Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε αυτό σαν κάτι παρόμοιο με το αμερικανικό μοντέλο που έχουμε την ε, ομοσπονδιακή κυβέρνηση όπου πάνω από το 50% των δαπανών το αποφασίζει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Αυτό αποκλείεται να γίνει στην Ευρώπη. Εμείς θα έχουμε μια πολύ πιο περιορισμένη ομοσπονδιακή διάσταση, ένα μικρό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που θα είναι το πολύ 2 με 3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Το οποίο δεν είναι λίγο. Το ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι το 2-3% του ΑΕΠ μπορεί να μας εξασφαλίσει μια καλά λειτουργούσα νομισματική ένωση. Γιατί τα δημοσιονομικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μπορεί να αντιμετωπιστούν με ένα προπολογισμό 2 με 3% του ΑΕΠ τη Ευρωζώνη. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μα όπου εξηγώ γιατί επαρκεί αυτό το ποσοστό. Ευχαριστώ Στεφάν. Θέλω να, να απαντήσω καταρχά και εγώ στου Γάλλου βουλευτέ. Κύριε Μάλκ, μιλήσατε για τι εκλογέ ε, του κυρίου Ολόντ που άλλαξε τη συνένεση στην Ευρώπη. Αναμφιβόλως αλλά αυτό δεν λύνει το βασικό πρόβλημα. Αλλάζουμε τη συνένεση, αλλά τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Σολάντ ίσως κατάφερε να αλλάξει την άποψη της κυρίας Μέρκελ εν μέρη, αλλά σε εσωτερικό επίπεδο στη Γαλλία κάποιοι θα χάσουν ούτως ή άλλως. Γιατί τελικά η ανάπτυξη που είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο κύριος Σολάντ δεν έχει επιτευχθεί. Πώς θα υλοποιηθεί. Η Γαλλία λοιπόν δεν είναι το καλό παράδειγμα. Η Ελλάδα είναι το σωστό παράδειγμα. Όπου είχαμε εκλογικά αποτελέσματα που δεν άρεσαν στους Ευρωπαίους. Τελικά διαλύσαμε το λαό και εκλέξαμε έναν άλλο λαό. Το θέμα μπορεί να τεθεί αύριο μεθαύριο στην Ιταλία. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που μπαίνει σήμερα. Το βασικό ερώτημα που μπαίνει σήμερα. Ο κύριος Καρές έκανε μια διάκριση, μια παρατήρηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρθηκε στην Ομοσπονδία στην Αμερική, στο Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Σύστημα, καθώς επίσης και στον Ομοσπονδιακό Έλεγχο ο οποίος γίνεται ανεξάρτητα από τον τοπικό έλεγχο. Μολονότι οι ομοσπονδιακές τάσεις στην Ευρώπη εξελίσσονται διαφορετικά και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ε, οι περισσότεροι είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας γιατί τελικά σε τι καταλήγει, σε έναν έλεγχο του τοπικού επίπεδου. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τον γερμανικό ομοσπονδιασμό, της ε, Βαβαρίας για παράδειγμα, όπου το τοπικό έπρεπε να ελέγχει το ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι το αμερικανικό σύστημα ομοσπονδίας βρίσκεται πραγματικά πιο κοντά σε αυτό που θα έλεγα δημοκρατικό μοντέλο. Για ποιο λόγο. Γιατί ο έλεγχος γίνεται σε σχέση με τον πολίτη που επηρεάζεται από μια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν ο Ιρλανδός βουλευτής είπε ότι θα πρέπει να φέρουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο κοντά στον πολίτη, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ θα το ήθελα, αλλά παραμένει έμεσο. Και αυτό τελικά βλέπουμε. Και αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η αντίφαση την οποία σας εξήγησα. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν μπορεί το μοντέλο αυτό να λειτουργήσει. Χρειάζεται ένας άμεσος έλεγχος από τους πολίτες, γιατί οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν, λαμβάνουν τις επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών, όχι τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ως κυρίαρχος πολίτης, εγώ θέλω να μπορώ να επιλέγω και δεν μπορώ να το κάνω αυτό όσοι εκλογές γίνονται εν μέρη. Στα γερμανικά θα απαντήσω στη συνέχεια. Τώρα για την ε, κοινή γνώμη. Ποια είναι η κοινή γνώμη, από πού προκύπτει η κοινή γνώμη. Αυτά τα ερωτήματα τα θέτει και, η... και το Συνταγματικό Δικαστήριο. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη, άρα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μα είναι λάθος αυτό. Εφόσον υπάρχει άμεσος έλεγχος των πολιτών επί των πολιτικών αποφάσεων, δημιουργείται κοινή γνώμη. Οι πολιτικοί όπως εσείς που είστε εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να δημιουργήσουν πλειοψηφίες. Για να δημιουργήσουν πλειοψηφίες περνάνε από τη μία χώρα στην άλλη για να κάνουν συζήτηση ούτως ώστε να υπάρξει συνένεση για τις επιλογές που προτείνουν. Αυτό δημιουργεί κοινή γνώμη. Αυτή είναι η κοινή γνώμη. Είναι επίπτωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Βεβαίως, είπαμε «Α, κάποιος τρελάθηκε όταν άκουσε τη λέξη δημοκρατία». Republic. Δημοκρατία σημαίνει «res publica», κοινό αγαθό. Είναι το κοινό αγαθό που κατέχουμε και είναι η διοκτησία δικό μας, των πολιτών, όχι των κυβερνήσεων. Εμείς είμαστε διοκτήτες αυτού του κοινού αγαθού. Και ως ιδιοκτήτες θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα απόφασης. Αλλά ευρωπαϊκή δημοκρατία λοιπόν σημαίνει αυτός ο μικρός αλλά σημαντικός τομέας του res publica που μας επηρεάζει όλους. Αυτό το μικρό αλλά σημαντικό στρώμα. Είναι διεθνής δημοκρατία. Πρέπει να το συζητήσουμε, να αναπτύξουμε ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις εθνικές δημοκρατίες με την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αλλά ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Κόβουμε σε οριζόντια τμήματα την Ευρώπη, όχι κάθετα όχι κάθετα όπου να συνδέονται όλα, που να έχουμε από το χαμηλότερο επίπεδο στη Βαβαρία τη δυνατότητα συζήτηση για το υψηλότερο στην Ευρώπη. Οπότε είμαι πλήρω υπέρ μια σταδιακή προσέγγιση, βήμα το βήμα. Βεβαίω, α αρχίσουμε σήμερα εδώ τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Αλλά αυτό που δεν θέλω είναι βήμα με βήμα να οδεύουμε όλο και περισσότερο προς αδίέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χάνιγκαν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρέπει καταρχάς να πω ότι ακούσαμε κάποιες εξαιρετικές παρεμβάσεις ε, σήμερα το απόγευμα. Ένα ηγητής συνόψε τη ζήτηση πάρα πολύ καλά όταν είπε ότι ζούμε σε μία περίοδο άμεσων αντιδράσεων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ γρήγορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξαιτία λοιπόν τη σημασία για την εφαρμογή άμεσα των αποφάσεων αυτών, πολύ συχνά οι εθνικοί βουλευτέ δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να συμμετέχουν στι διαδικασίε διαβούλευση. Και τελικά, είναι οι εθνικοί αυτοί βουλευτέ που πρέπει να λογοδοτήσουν στη συνέχεια στου πολίτε του. Πρέπει να πάνε, να του εξηγήσουν, να επεραμεινθούν συγκεκριμένων πολιτικών και το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι δεν έχουν συμμετάσχει πάρα πολύ στην διαδικασία και θεωρώ ότι η διάσκεψη των Προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Κύπρο θα ασχοληθεί και με το ζήτημα αυτό. Ένα ομιλητή με ρώτησε ποιο θα είναι το πόρισμα τη ε, συνεδρία αυτή. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το άρθρο 13, δηλαδή ποιε θα πρέπει να είναι οι αρμοδιότητε και οι ευθύνε των Εθνικών Κοινοβουλίων σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώ ορίζονται αυτέ στο άρθρο 13 και τι είδου επίβλεψη εμεί μπορούμε να έχουμε ω εθνικοί βουλευτέ. Αυτό πραγματικά ελπίζω ότι θα είναι το αποτέλεσμα τη συνεδρία στην Κύπρο. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος του ΕΛΚΟ πρώτος ομιλητής και θα ακούσουμε επίσης και την Ελίζα Φερέιρα. Φέιο. Και η Ελίζα Φεραίρα συνέχεια θα μας μιλήσει συγκεκριμένα για την έκθεσή της για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο κύριος Φέιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας πραγματικά όλους τους συναδέλφους, μέλη του, των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι Ευρωβουλευτής. Πρώτη φορά συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο παρελθόν υπήρξα βουλευτής του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η πρώτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορώ να πραγματικά καταλάβω και τι δύο πλευρέ τι οποίε συζητάμε σήμερα. Το πρώτο ζήτημα που θέλω να θίξω είναι η σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεί πραγματικά μια γέφυρα ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδίω, ε, μάλλον επισημοποιείται κατά κάποιο τρόπο αυτή η σχέση. Ω απόρρια τη όλη εργασία που έχει γίνει στα πλαίσια του Six προσπαθήσαμε να δούμε πώ από πολιτική πλευρά μπορούμε να επιβλέψουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διάφορε εναλλακτικέ που μπροστά τη ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σα πω ότι μιλώ εξ ονόματο του κυρίου Γκοζέ, ο οποίο ήταν σκιώδη ηγητή εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, όσον αφορά την έκθεση τη κυρία Φερέιρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα ήθελα λοιπόν να σα πω ότι ε, Δύο από τις πιο βασικές έννοιες ε, της διασύνδεσης ε, Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση, ζήτημα το οποίο καλύψαμε διεξοδικά σήμερα και ζήτημα που αποτελεί τμήμα των ε, πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνουν οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξετάζοντας την τήση επισκόπηση ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει καταρχάς να πω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να υποβάλει κάποιες ε, ιδέες που θα επηρεάσουν τελικά τα κράτη-μέλη και επί των οποίων θα πρέπει να αποφανθεί το Συμβούλιο, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι ιδέες αυτές προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, ότι επιτρέπουν στην οικονομία να λειτουργήσει ομαλά, ότι καταπολεμείται η ανεργία, ότι εξυγχρονίζονται οι δημόσιες διοικήσεις και ότι εν τέλει αυξάνεται η πολιτική επιτήρηση, η πολιτική εποπτεία όλων αυτών των ζητημάτων. Στα ζητήματα αυτά ουσιαστικά θα πρέπει να αναφέρεται η αιτήσια επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη. Προκειμένου εμείς να καταφέρουμε τώρα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, προκειμένου να αυξηθούμε, να αναπτυχθούμε οικονομικά, θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας. Και αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρχει πραγματικά μία δημοσιονομική πειθαρχία, αν υπάρχει μεταξύ μόνο καλύτερη εμπιστοσύνη και αν προχωρήσουμε σε απαραίτητε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Η Ευρώπη έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές αυτές, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι σε πολλές χώρες ακολουθούσαμε λαθασμένα οικονομικά μοντέλα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πιστεύω ότι έχει έρθει πλέον ο χρόνος για να αντιμετωπίσουμε σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Προέρχομαι, όπως σας είπα, από την Πορτογαλία. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα καλό καθεστώς δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για πολλούς πολίτες να αποδεχθούν τέτοιες αποφάσεις. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι αντιμετωπίζουμε απλώς αυτή τη στιγμή μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το παρόν μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να περάσουμε από το στάδιο αυτό, από τη φάση αυτή, για να ταινίσουμε έπειτα ένα πιο θετικό μέλλον θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους. Αυτό γίνεται όλο και περισσότερο ε, έκδηλο. Χρειαζόμαστε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις Θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίε του κάθε κράτου μέλου, το είπε αυτό και όλοι Ρεν, ο Επίτροπο, και θα πρέπει όμω να υπάρχει και ένα υψηλό επίπεδο συνένεση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τον, μέσω των συναντήσεων εθνικών και ευρωπαϊκών βουλευτών, εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών, με συγχωρείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως υπόθηκε, να καταφέρουμε να έρθουμε πιο κοντά στους εκλογείς μας. Προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο όμως, θα πρέπει να αρχίσουμε να τους μιλάμε για πράγματα τα οποία τελικά επηρεάζουν τη ζωή τους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα πρέπει τελικά να καταφέρουμε μεταξύ μόνο να συμφωνήσουμε για όλα αυτά τα σημεία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Ελίζα έχει το λόγο για να ολοκληρώσει τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πιστεύω ότι πραγματικά η συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Κατά την άποψή μου, ουσιαστικά αναφερθήκαμε σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη διανύουμε μια δύσκολη φάση, μια επικίνδυνη φάση, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να ταινίζουμε το μέλλον τελικά, προκειμένου να καταφέρουμε να βγούμε από τη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα αυτό. και πιστεύω ότι γίνανε πάρα πολύ κέρυες παρεμβάσεις προς αυτό. Η Ευρώπη διανύει μία περίοδο όπου βλέπουμε τελικά ότι έχει μείνει πίσω, ή λείπεται. βλέπουμε ότι οι υπόλοιπε χώρες προχωρούν πολύ περισσότερο στον τομέα της παγκοσμιοποίησης και βλέπουμε επίσης ότι διανύουμε μία περίοδο όπου ουσιαστικά έχει κλονιστεί και έχει δοκιμαστεί, θα έλεγα πολύ, το νέο νόμισμα. Πρέπει να περάσουμε όμω πλέον την περίοδο αυτή. Πρέπει να αποκομίσουμε σημαντικά διδάγματα από την περίοδο αυτή και να συνεχίσουμε σε μια μελλοντική πλέον περίοδο. Σίγουρα μέσω πολύ δύσκολων κρίσεων που κλώνησαν πάρα πολλές κοινωνίες, πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα. Είδαμε πόσο σοβαρές ήταν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες που υπήρχαν ανάμεσα στα κράτη-μέλη πόσο σημαντικό να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες αυτές και πόσο σημαντικό να καταφέρουμε να πάρουμε τι σωστές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάθαμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε πέρα από το νέο νόμισμα και να καταφέρουμε να θεσπίσουμε τελικά μια καλύτερη θεσμική αρχιτεκτονική η οποία να στηρίζει αυτό το ευρωπαϊκό νόμισμα. Η ευρωπαϊκή αυτή διάρθρωση ναι είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές οι οποίες πιστεύω ότι πραγματικά βελτιώνουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών. Στο Συμβούλιο των Υπουργών μάλιστα έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα ο ρόλος του ΕΚΟΦΗΝ και έχει ενισχυθεί επίσης και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά όπως είπαν και πολλοί ομιλητές, η κρίση έχει τονίσει την ανάγκη για άμεσες ταχείες απαντήσεις για άμεση λήψη μέτρων. Πράγμα το οποίο έκανε τελικά το ευρωπαϊκό επίπεδο πολύ πιο παρεμβατικό στο εθνικό, στο τοπικό επίπεδο, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και οδήγησε σε μία μείωση κυριαρχία για ορισμένα κράτη-μέλη και το ζήτημα αυτό το θίξαμε σήμερα το απόγευμα. Τίθε λοιπόν το ζήτημα τη νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται και το πώ θα καταφέρουμε τελικά να συμφιλιώσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα με τα συμφέροντα μεμονωμένων κρατών μελών. Και αυτό το ζήτημα απομένει να το επιλύσουμε. Θα τόνιζα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιδέα που ακούστηκε της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Πολύ ωραίο το μήνυμα, πολύ ωραία εικόνα που κρύβεται πίσω από την έννοια αυτή. Ουσιαστικά πώς θα καταφέρναμε να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο λοιπόν η ιδέα αυτή. Άκουσε επίσης τα όσα είπε ο καθηγητής Βόλφ, τα οποία ζητήματα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία ευρωζώνη, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα προπολογισμό για την ευρωζώνη αυτή. Πώς μπορούμε να εξορροπήσουμε καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη και σε αυτές που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης. Πώς μπορούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των μικροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνη. Έρχομαι κατά αυτόν τον τρόπο στο six-pack. Πιστεύω λοιπόν ότι βασιζόμενοι στο six-pack θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αποφάσεις οι οποίες να λειτουργούν προς όφελος της Ευρώπης. Πρέπει να πετύχουμε μια εξορρόπηση. Κάπου θα νικήσουμε και κάπου θα ετηθούμε. Αλλά παντού θα πρέπει να έχουμε ως κοινό γνώμονα το κοινό καλό δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε, στην κατάσταση εκείνη όπου κάποιοι τελικά θα βγουν απολύτω νικημένοι από το παιχνίδι αυτό και ορισμένοι θα Αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία τελευταία παρατήρηση. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι επειδή έχουμε και την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την έκθεση της ετήσιας επισκόπης για την οικονομική ανάπτυξη. Έχω συνεργαστεί με τους αδέλφους μου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και μαζί τους τους το έχω πει και το λέω και σε εσά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος. Ελπίζω λοιπόν ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα, από το ΕΛΚ θα φροντίσουν να καταλήξουμε σε κάποιους συμβασμούς. Δεν μπορούμε μέσω της αναδίπλωσης να επιλύσουμε τα προβλήματα. Αντίθετα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πιο εντατική συνεργασία και διαβούλευση. Πιστεύω λοιπόν ότι όσον αφορά το 2013 μπορούμε πραγματικά να ξεκινήσουμε τώρα την εργασία για να αυξήσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένους συμβασμούς και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και σημαντικές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν καταλήκλειδη θα έλεγα ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πιο ισορροπημένη μέθοδο συνεργασίας με τους εθνικούς βουλευτές. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι θα αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο και τι θα αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό η κοινοτική μέθοδος να ενισχυθεί. Γιατί η διακυβερνητική μέθοδος ουσιαστικά έχει κάποιες αδυναμίες οι οποίες είναι πλέον σαφείς. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιστρέψουμε σε μια τέτοια μέθοδο. Πρέπει ανταυτού να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στην κοινοτική μέθοδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πάρα πολύ καλή διασύνδεση με τα εθνικά κοινοβούλια. Όπως το είπε και ο Επίτροπος Ολιρέν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι εθνικοί βουλευτές ότι μπορούν να έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όποτε το επιθυμούν και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συνεχής διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες αρμοδιότητες του Eurogroup που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο, χωρίς όμως να θέτουμε εν κινδύνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με την προεδόρο μας, την κυρία Μπόλς. Όντως βρισκόμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Και να απόκειται σε εμά να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα διέξοδα τα οποία έχουν προκύψει, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή και να δώσουμε νέα όθηση στην Ευρώπη. Και να μην δίνουμε απλώ τη σύμφωνη γνώμη μα σε κάποιε προτάσει. Αν δεν καταφέρουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί με ένα ισορροπημένο τρόπο, τότε θα χάσουμε όλοι μαζί από κοινού. Πιστεύω ότι μπορούμε να αποκομίσουμε πολλά μαθήματα ακόμα και από τεφιστάμενα εμπόδια και θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να αγγλίμουμε διδάγματα και στη συνέχεια να συζητάμε μεταξύ μας και να εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε μάλλον, για το κοινό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ μπορώ να πω ότι έχω μάθει πολλά εξαιρετικά πράγματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τελειώσαμε ακριβώς την ώρα μας. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα δύο-τριών λεπτών για να αλλάξουν οι ομιλητές και θα ξαναρχίσουμε για το δεύτερο τμήμα. Όσοι είχαν συμπληρώσει κάρτες ε, λέγοντας ότι θέλουν να μιλήσουν και στα δύο τμήματα. Τα έχω κρατήσει. Ήδη έχουμε ένα αρκετά σημαντικό κατάλογο, αρκετά, αρκετά, ε, τέτοιες, αρκετά τέτοια έντυπα, αλλά παρακαλώ όποιοι άλλοι θα ήθελαν ε, να συμπληρώσουν και εκείνοι. Σε δύο λεπτά λοιπόν ξαναρχίζουμε. Okay, if we take our seats ready for the second... Παρακαλώ, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης μας σε λίγο. Λοιπόν, για να καλύψω το χρόνο μέχρι να έρθετε όλοι. Το δεύτερο τμήμα είναι ως, έχει ως τίτλο το ερώτημα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ε, είναι η πολιτική μας ε, βασισμένη στην ε, λιτότητα ή στην ανάπτυξη γιατί ορισμένοι λένε ότι είναι υπερβολικά στενό το πλαίσιο που έχει για να καθορίσει την πολιτική μας ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο πώς θα μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και ε, απασχόληση η συζήτηση αυστηρό, λιτότητα έναντι απασχόλησης μπορεί να ξαναγίνει με νέο ε, οπτικό κέντρο μετά τη συζήτηση για τους προπλησιαστές και πιστεύουμε ότι οι πολιτικές μας θα αποδώσουν μόνο μέσω πρόθεσμα ή χρειάζεται ριζική επανεξέταση της πολιτικής μας για να υπάρξουν μαζικές δημόσιες επενδύσεις. Καλωσορίζω τον Hans Werner Zinn που είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου IFO για, οικονομική, ε, για οικονομικές μελέτες και τον κύριο Τίμπο που είναι διευθυντής ε, του Γαλλικού ε, Κέντρου Μελετών FCA για θέματα αναλύσεων και προβλέψεων. Έχουν διαφορετικές απόψεις για τα θέματα που έχουμε θέσει οι ομιλητές. Ελπίζω αυτό να οδηγήσει σε έντονο και επικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Στόχος μας είναι οι ομιλητές μας να προκαλέσουν συζήτηση και όχι απλώς να απευθυνθούν ε, στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή αποδοχής απόψεων που υπάρχει ανάμεσά μας. Δίνω λοιπόν πρώτα απ' όλα το λόγο στον Hans Werner Zinn. Δέκα λεπτά παρακαλώ, να ο χρόνος σας. Κύρια Μπάουλς, διακεκριμένη παρεπρισκόμενη, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω. Λιτότητα ή ανάπτυξη. Είναι λάθος ερώτημα διότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσω της λιτότητας. Η ανάπτυξη μέσω πολιτικής τόνωσης της ζήτησης ε, και ενσιανών πολιτικών δηλαδή θα βελτιώσει κάποιες ε, καταστάσεις αλλά δεν θα προκαλέσει ανάπτυξη. Πρέπει να βελτιώσουμε τι δυνατότητε των οικονομιών, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Και εδώ έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη. Όταν αναγγέλθηκε το 1995 το ευρώ, όπω ξέρετε, προσπάθησε να προκαλέσει σύγκληση των επιτοκίων. Αυτό έδωσε το μήνυμα στους επενδυτές ότι παντού ήταν ασφαλεί οι επενδύσει του. Μικρέ λοιπόν διαφορέ στα επιτόκια σήμαιναν μεγάλε μεταφορέ επενδύσεων από τον βορρά στον νότο. Καταρχήν αυτό ήταν εποφελέ, διότι βοήθησε την μείωση των ε, ανισοτήτων εισοδημάτων. Αλλά στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαμε αυτό σήμαινε πολλές αυξήσεις ε, για τις ε, Απολαβέ των δημοσίων υπαλλήλων. Στην Ισπανία είδαμε την φούσκα των ακινήτων και οι δύο αυτές προσεγγίσεις είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Υπήρξε μια τεράστια τεχνητή ανάπτυξη της οικονομίας, προκάλεσε και πραγματική αύξηση, αλλά προκάλεσε και πολύ πληθωρισμό. Ίσως να έχετε το έγγραφο μπροστά σας, όπου έχω συνοψίσει μερικά σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Εκεί βλέπετε τα πρώτα στοιχεία αυτή η τεράστια άξη των τιμών από την συνάντηση κορυφής στη Μαδρίτη όπου πραγματικά αναγγέλθηκε η δημιουργία του ευρώ βλέπουμε μια αύξηση του 67% και όλες οι, στην Ελλάδα και όλες οι άλλες χώρες της κρίσης είχαν μεγάλη αύξηση ενώ στη Γερμανία έχουμε μόνο 9%. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες χώρες, οι χώρες που σήμερα βρίσκονται σε κρίση ανατίμησαν μέσω του ευρώ την οικονομία τους σε πραγματικούς όρους. Ενώ άλλες υποτίμησαν την οικονομία τους. Αυτή η άνα και υποτίμηση συνολικά μας έχει οδηγήσει σε λάθος τιμές. Αυτές είναι το πρόβλημα. Ορισμένες χώρες έχουν γίνει πολύ ακριβές για να είναι ανταγωνιστικές και θα χρειαζόμασταν μία αναπροσαρμογή των ισοτιμιών για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί έχουμε ένα νόμισμα. Αν πάρουμε τις έξι χώρες που ε, πλήττονται μαζί από την κρίση, συνολικά ανατίμησαν την οικονομία τους από το 1995, αν συμπεριλάβουμε και την περίοδο ανοιχτής προσαρμογής των ισοτιμιών, ανατίμησαν κατά 30%. Τι δυνατότητε του σε σχέση με τους εμπορικούς τους εταίρους. Ενώ στη Γερμανία, αντίθετα, υπήρξε υποτίμηση κατά 22%. Αυτές είναι τεράστιες διαφορές. Εξηγούν γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Ορισμένες χώρες έχουν βαλτώσει τώρα στο πολύ υψηλό επίπεδο τιμών τους και δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα μέχρι το 2007, γιατί τα τεράστια ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών χρηματοδοτούνται από τις χρηματαγορές. Αλλά όταν ήρθε η κρίση στην Ευρώπη, το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν ήθελε να χρηματοδοτεί πλέον αυτά τα ελλείμματα. Τότε βεβαίως ε, πήρε μπρο ε, το... ο μηχανισμός για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων και ο δευτερογενής ε, τομέας οι βόρειες τράπεζες αναγκάστηκαν να αγοράσουν τα νότια ομόλογα. Στην ουσία δηλαδή υπήρξε αυτή η δημόσια ροή, η ροή μάλλον δημοσίων αγορών αντικατέστησε τις ε, ροές των ιδιωτικών αγορών, αλλά μακροπρόθεσμα αυτή η λύση δεν αποδίδει. Οι χώρες που έχουν γίνει πολύ ακριβές πρέπει να ξαναγίνουν φτηνότερες. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στην πρώτερη κατάσταση ένα παλιό ρολόι. Όπως ξέρετε, πολλές φορές ε, ε, τα χέρια του ε, πηγαίνουν μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Πώς λοιπόν θα το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω προγραμμάτων αποπληθωρισμού και λιτότητας, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσουν, αυτά τα προγράμματα μπορεί να δημιουργήσουν τρομερές ρήξεις στην κοινωνία. Βεβαίως, ξέρουμε τι έγινε στη Γερμανία κατά την περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Η Γερμανία είχε γίνει πιο ακριβή σε σχέση με τους ε, εμπορικούς της εταίρους επειδή βέβαια υπήρχαν σταθερές ε, ισοτιμίες στη Γερμανία έναντι του, δολαρί, ε, έναντι χρυσού ενώ σε άλλες χώρες δεν υπήρχε κάτι τέτοιο προσπάθησε η Γερμανία να μειώσει τους μισθούς οι μισθοί μειώθηκαν σε τέσσερα χρόνια κατά 28% και οι τιμές κατά 23%. Αυτός ήταν ε, ο στόχος της πολιτικής, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουμε στα πρόθυρα ε, του εμφυλίου πολέμου και τελικά αυτό που προέκυψε το 1933 ήταν χειρότερο από εμφύλιος πόλεμος. Ο Κέιντς παρατηρώντας αυτά τα φαινόμενα θεώρησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αναπροσαρμογή μέσω μειώσεων μισθών και τιμών και ο Φρίντμαν ο αντίπαλός του για διάφορα θέματα συμφωνεί σε αυτό. Υπάρχει ευρεία αποδοχή μεταξύ των οικονομολόγων ότι αυτή η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω προγραμμάτων λιτότητας. Ωστόσο, αν θέλουμε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των χωρών, δεν υπάρχει άλλη ανακτική. λύση. Πρέπει να αλλάξουν οι σχετικές τιμές. Πόσο πρέπει να αλλάξουν. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Goldman Sachs, που διαρκεί ακόμη στην περσινή τους εκδοχή, αλλά και σε αυτή που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθούν να καθορίσουν κατά πόσο πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε σχέση με τον ε, μέσο όρο της Ευρωζώνης για να γίνουν ανταγωνιστικές κάποιες χώρες. Και να τα στοιχεία. Για την Ισπανία είναι 30%, για τη Γαλλία 20%, για την Ελλάδα και την Πορτογαλία 30% επίσης. Ή μια άλλη σύγκριση Ελλάδα με Τουρκία που έχουν ε, παρόμοιες συνθήκες. Η Ελλάδα είναι 64% πιο ακριβή από την ε, Τουρκία. Θα χρειαζόταν λοιπόν για να ανταγωνιστεί την Τουρκία υποτίμηση 39%. Τι ποσοστό υποτίμηση έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα στη σελίδα 10 που δείχνει την πραγματική ισοτιμία όπως την καθορίζει η Eurostat αυτό είναι το αποπληθωρισμένο ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Εδώ θα δείτε ότι πολύ λίγα έχουν γίνει. Οι τιμές κατά την κρίση ακολούθησαν ε, παράλληλη πορεία. Οπότε η αναγκαία υποτίμηση στις χώρες που, είχε γίνει πολύ, που είχαν γίνει πολύ ακριβές δεν συνέβη. Και δεξιά βλέπετε τις εκτιμήσεις ε, της Goldman Sachs για το πόση υποτίμηση πρέπει να γίνει σε αυτές τις χώρες και πόση ανατίμηση στη Γερμανία. Η Γερμανία θα πρέπει να έχει πληθωρισμό 20% σε σχέση με το μέσο όρο και η Γαλλία να υποτιμήσει κατά 20% σε σχέση με το μέσο όρο. Αυτές είναι τεράστιες αλλαγές. Δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να γίνει. Είναι δυνατόν, όπως σας είπα αρχικά, η Γερμανία σε 13 χρόνια υποτίμησε κατά 22% έχοντας χαμηλότερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες. Αλλά φυσικά δεν ήταν ευχάριστο, σημαίνει τεράστια ανεργία. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να κάνει οδυνηρές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις Σρόντερ, για παράδειγμα, σήμαιναν ότι ε, πολλοί Γερμανοί έχασαν επιδόματα για να μειωθούν οι απολαβές τους και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό που έκανε η Γερμανία πριν από 10 χρόνια είναι η διαδικασία που χρειαζόμαστε τώρα στις χώρες που έχουν γίνει πολύ ακριβές. Ε, θα μπορέσουν να το κάνουν εντό της Ευρωζώνη όλε αυτέ οι χώρε. Ε, προσυζήτηση. Εγώ αμφιβάλλω. Νομίζω ότι ορισμένες έχουν απομακρυνθεί υπερβολικά από το σημείο ισορροπίας για να είναι σε θέση όντως να αντέξουν τόσο μακρά περίοδο στασιμότητας που θα είναι αναγκαία. Αλλά δεν θέλω να θέσω αυτό προς συζήτηση. Φυσικά μπορεί να γίνει και χωρίς μειώσεις τιμών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε χωρίς περικοπές τιμών. Αν υποθέσουμε ότι οι τιμές στην Ισπανία θα παραμείνουν σταθερές, τότε για να επιτύχει την αναγκαία αναπροσαρμογή εντός μιας δεκαετίας έχω κάνει τις, ε, τους υπολογισμούς εδώ θα έπρεπε κατά μέσο όρο η Ευρωζώνη να έχει πληθωρισμό 3,6% και η Γερμανία να έχει πληθωρισμό 5% και μετά από μια δεκαετία στασιμότητας για την Ισπανία θα έχει ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της δεν είναι αυτή η αυστηρή λιτότητα που θα μειώσει τις τιμές, αλλά και αυτό δεν θα είναι ευχάριστο. Δεν έχουμε άλλη λύση. Έχει παγιδευτεί η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση από όπου από οικονομικής πλευράς δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Παρά τους ε, κυριακάτικους λόγους των πολιτικών το πρόβλημα στην Ευρώπη παραμένει. Δεν μπορούμε με ευσεβείς πόθους να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρξουν σκληρά μέτρα. Είτε λοιπόν η Ευρωζώνη θα μπορέσει να επιτύχει αυτές τις αναπροσαρμογές μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια, είτε δεν θα επιζήσει το ευρώ. Δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη μου άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Δεν υπάρχουν. Όσο νωρίτερα το καταλάβουμε τόσο καλύτερα. Πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης και ενσιανές θα βοηθήσουν προσωρινά τεχνητά θα δημιουργηθεί η ζήτηση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά αλλά είναι σαν αναλγητικό απλώς αναβάλει την αναγκαία θεραπεία που χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και τέλος πρέπει οπωσδήποτε ο Βοράς και ο Πυρήνας να ανατιμήσουν την οικονομία τους Πώς θα το κάνουν αυτό. Ορισμένοι λένε ας αυξήσουμε τους μισθούς. Αυτό είναι ανόητο. Αν τεχνητά αυξήσουμε τους μισθούς, δημιουργείται στάσιμο πληθωρισμό. Το θέμα είναι πώς θα αυξήσεις τους μισθούς. Πρέπει να τους αυξήσεις μέσω αύξησης της ζήτησης. Ζήτηση για εργασία, ζήτησης, αύξησης της ζήτησης. Αυξάνοντας απλώς τους μισθούς δημιουργείς ανεργία, στασιμότητα της οικονομίας, μείωση των εισαγωγών και η κατάσταση θα γίνει χειρότερη για τις νότιες χώρες. Πώς θα αυξηθεί η ζήτηση μόνο μέσω των δυνάμεων της αγοράς. Οι δυνάμεις της αγοράς στην κρίση αυτή δεν θέλουν να πάνε πια στη Νότια Ευρώπη όσο ήθελαν. Όπως ξέρετε, τα γερμανικά κεφάλαια εξήγονται μέσω του τραπεζικού τομέα στη Νότια Ευρώπη. Τα κεφάλαια δεν θέλουν πια να πάνε στην Νότια Ευρώπη. Φυσικά προσπαθούμε να τους πρόξουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν επαρκεί. Όσο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο δεν θα υπάρξει ένα προσαρμογή. Πρέπει να αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει. Τότε θα υπάρξει μια αύξηση της οικονομίας στο βορρά που είναι αναγκαία για να μειώσει πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών του βορρά και έτσι ο Νότος θα αποκτήσει περισσότερα επίσης. Θα αποκτήσει λιγότερο έλλειμμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι πρέπει να στείλουμε τις οικονομίες του Βορρά στο Νότο μέσω δημοσίων μέτρων στήριξης και την ίδια στιγμή να ζητάμε να μειωθούν οι ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών αλλαγών θα ήταν παράλογο κάτι τέτοιο, γιατί επιχειρούμε δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ξαβιέ Τεμπό θα μας κάνει μια άλλη παρουσίαση τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω γαλλικά, αν μου επιτρέπετε. Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα και θα είναι πολύ πιο ευχάριστο για σας που δεν θα ακούτε τα άσχημά μου αγγλικά. Έχω κάποιες αγγλικές διαφάνειες οι οποίες θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να παρακολουθήσετε αυτά που θα σας πω. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να σας εμπιστήσω την προσοχή είναι ότι σήμερα στην Ευρώπη, σε ορισμένους, όχι σε όλους, και ο καθηγητής ε, ΣΥΝ δεν ανήκει σε αυτούς, υπάρχουν ε, κάποιοι που βλέπουν ότι βελτιώνεται η κατάσταση, ότι υπάρχουν σημάδια. Υπάρχουν κάποια σημάδια. Το πρώτο σημάδι είναι ότι σταματάμε να μιλάμε για τη διάλυση του ευρώ. Ένα δεύτερο από το σημάδι είναι ότι η κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι σε φάση σταθεροποίησης. Ίσως διαβάσατε στον τύπο ότι πρόσφατα οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, πρόωρα επιστρέφουν τα δάνεια που του έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεσοπρόθεσμα. Αυτό είναι σημάδι ότι έχουν εκ νέου ρευστότητα οι τράπεζες ε, και υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών. Υπάρχει ένα άλλο σημάδι επίσης παρότι είμαστε σε ψηλά επίπεδα, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν πρόσβαση πιο εύκολα στις ε, αγορές. Και ο φόβος ότι θα στερέψει το χρήμα από τις αγορές και ότι δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το χρέος τους, αρχίζει να εκλείπει. Θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά τα θετικά στοιχεία είναι ένα φως στο βάθος του τούνελ, που μας λέει ότι περάσαμε από κάποιες δοκιμασίες, αποφύγαμε το χειρότερο και τελικά βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση επιτέλους. Θέλω να σας πω ότι το φως αυτό στο βάθος του τούνελ μπορεί να είναι το φως του τρένου που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, μια καταστροφή που έρχεται που απειλεί τις οικονομίες μας και όχι η ελπίδα ότι θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είδαμε πολλά τρένα να έρχονται κατά μέτωπα τι γίνεται με αυτό το φως τώρα που βλέπουμε. Μπορούμε να πούμε ότι για ακόμα μία χρονιά, για την πέμπτη συναπτή χρονιά, η Ευρωζώνη έχει αρνητική ανάπτυξη. Είχαμε, μετά, από, είχαμε διάφορα χρόνια μετά το 2008 ε, χαμηλή ανάπτυξη ή αρνητική ανάπτυξη. Η ανεργία έφτασε στην Ευρωζώνη σε επίπεδα ρεκόρ. Σε ορισμένε χώρες έφτασε σε επίπεδα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Στην Ισπανία, α πούμε, η ανεργία ξεπερνάει το 26%. 26% είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Το 1 τέταρτο του ενεργού πληθυσμού δηλαδή δεν βρίσκει δουλειά. Είναι ποσοστά που είχαμε δει στο μεγάλο κράχ της ΗΠΑ, Πολιτείες, δεκαετία του 30. Είναι ποσοστά ανεργίας που παραπέμπουν σε καταστάσεις που δεν είναι καταστάσεις ύφεση, αλλά βαθύτατη ύφεση. Αυτό ζει αυτή τη στιγμή η Ισπανία. Όλη αυτή η κρίση επίση θα έχει επιπτώσει μακροπρόθεσμα. Οι επενδύσει, η προσπάθεια για την ανάπτυξη, οι δημόσιες επενδύσει, ε, οι επενδύσει στι υποδομέ, η εκπαίδευση και τα κονδύλια για όλα αυτά τα πράγματα κόβονται σε πολλές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικέ γενιές θα πρέπει να πληρώσουν Χωρί να μιλάμε για το θέμα του τι επίπτωση θα έχει αυτό στο περιβάλλον και στην οικολογία. Που κανονικά θα έπρεπε να μας αναγκάσει ήδη σήμερα να προωθήσουμε αυστηρές πολιτικές για να προετοιμαστούμε. Όμως, στη σημερινή κατάσταση ξεχνάμε το περιβάλλον, ξεχνάμε την οικολογία. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2013 είναι αρνητικές προβλέψεις. Γι' αυτό το φως απέναντι δεν είναι φως εξόδου. Οι προβλέψεις της Κομισιόν θα είναι αντίστοιχες με αυτές του, του ΟΣΑ, του Δουνουτού. Θα αναγγείλει και αυτή ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα είναι αρνητική, θα έχει αρνητικό πρόσημο. Κοιτάξτε τη δεύτερη διαφάνεια της παρουσίασής μου για να καταλάβουμε γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ενώ το ευρώ δεν θα διαλυθεί, ενώ σταθεροποιούνται οι Ευρωπαϊκέ τράπεζε, ενώ η Ισπανία και η Ιταλία εκ νέου μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από τις αγορές. Γιατί ακόμα μια χρονιά θα αντιμετωπίσουμε την ύφεση, την αύξηση τη ανεργία κτλ. Ο λόγος είναι απλός. Οι Ευρωπαϊκέ χώρε δεσμεύτηκαν από το 2010 και θα το συνεχίσουν αυτό το 2013 να προωθούν αυστηρότατα προγράμματα λιτότητες. Ορισμένες κασάνδρες λένε ότι βάλαμε τέτοια προγράμματα λιτότητας στα σκαριά, αλλά δεν τα εφαρμόσαμε. Μερικές φορές δεν εφαρμόσαμε σωστά, όντως, όπως προαναγγείλαμε. Αλλά όταν κοιτάξτε τον πίνακα στη δεύτερη διαφάνεια, τα νούμερα της μείωσης των διαρθρωτικών ελλημάτων, δηλαδή βγάζουμε τη συγκυρία από τα στοιχεία αυτά, όταν κοιτάμε τα νούμερα αυτά βλέπουμε ότι οι χώρες Ευρωζώνης δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν τεράστια προγράμματα λιτότητας. Και αυτά δεν είναι αναγγελίες ε, απλές. Έχουν προχωρήσει σε έργα. Ε, έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Το 2013 το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης θα συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα στην Ευρωζώνη θα έχουμε μια συρρήκνωση 1,4 του ΑΕΠ, του μέσα στο 2013 μόνο. Θα μου πείτε αυτό που σας είπε ο κύριος Ζήν, ο καθηγητής Ζήν, ότι χρειάζεται η λιτότητα για να περάσουμε συνεχεία στην ανάπτυξη. Να σε επιστήσω την προσοχή ότι χρειάζεται αυτή η λιτότητα για την ανάπτυξη και αυτό είναι μια ε, ιδέα, μια αντίληψη Υπάρχουν ε, εμπειρικά στοιχεία. Διαβάστε την έκθεση του EGES του 2013 που παρουσιάσαμε στο Κοινοβούλιο το Νοέμβριο. Διαβάστε τα κείμενα του Δουνουτού για αυτό το θέμα για να καταλάβετε ότι αυτό είναι παράδοξο. Είναι ένα παράδοξο. Γιατί σε φάσεις ύφεση, όταν έχουμε ψηλή ανεργία, όταν οι οικονομικοί φορείς λόγω των εισοδημάτων τους δεν μπορούν να ξοδέψουν ε, περισσότερα από ό,τι κερδίσουν, δεν μπορούν να προσφύγουν στους αγορές, είτε γιατί οι αγορές δεν λειτουργούν, είτε γιατί η κατάστασή τους ε, σημαίνει ότι αυτό θα έχουμε ρίξει. Ανεργία και οι χρηματαγορές δεν θέλουν να δανείσουν χρήμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που είχε πει ο Αμερικανός οικονομολόγος Ρομπέρ Μπαρό δεν λειτουργεί πια. Και βρισκόμαστε σε αυτό που είπε ο Κέινς τότε, ότι έχουμε ε, μία διαδοχική ύφεση. Σταματάω την κατανάλωση, μειώνω τα εισοδήματα και τα πράγματα επιδεινώνουν. Οι χρηματαγορές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτές τις συνέπειες. Έχουμε δηλαδή μία πολλαπλασιαστική επίπτωση αυτών των στοιχείων. Ε, και αυτοί οι πολλαπλασιαστικοί παράγοντες είναι πολύ πιο μεγάλοι όταν έχουμε ύφεση. Και έχουμε ύφεση. Όταν συρρυκνώνεται τον προπολογισμό, όταν έχετε δημοσιονομικές ε, περικοπές, αυξάνονται οι πολλαπλασιαστέ. Δείτε, δείτε τι γίνεται στην Ισπανία. Το 2009 είχαμε 9,3 ε, έλλειμμα του ΑΕΠ. Πολύ σημαντικό. Έκανε δημοσιονομικές προσαρμογές η Ισπανία τους βλέπετε στον πίνακα από τις αρχές του 2010 υπό διάφορες πιέσεις ε, του φόβου ότι θα στερέψει η χρηματοδότηση των αγορών προώθησε αυτές τις αλλαγές. Σήμερα το 2012, αυτή τη βδομάδα, η Ισπανική κυβέρνηση θα δημοσιεύσει την πρώτη εκτίμηση για το έλλειμμα του 2012 και θα είναι γύρω στο 8% του ΕΠ. Μετά από όλε αυτέ τις δημοσιονομικέ περικοπέ που έκανε η Ισπανία από το 2009, το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε το πολύ μείωση 1,3 του ελλείμματο. Αυτή είναι η φάση που ζει η Ισπανία, αυτή είναι η κατάσταση που ζει η Ισπανία. Το μόνο πράγμα που αυξάνει στην Ισπανία είναι η ανεργία. Δεν μειώνεται το έλλειμμα επαρκώ. Και όσο περισσότερο θα προσπαθήσει μέσω τη αλητότητα να μειώσει το έλλειμμα, η Ισπανία τόσο θα αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολυπλασιαστικό παράγοντα εδώ. Και αυτό, αυτή είναι η παγίδα της ύφεση. Όσο περισσότερο συρρυκνώνουμε την οικονομία, οικονομία, μειώνεται η εμπιστοσύνη στην Ισπανία. Η Ισπανία βρίσκεται σε μια όλο και πιο δύσκολη κατάσταση και μία από τις δυνατότητε να βγει από αυτή την κατάσταση θα είναι να πτωχεύσει. Όσο δεν έχει ανάπτυξη, ο κίνδυνος αυτός για πτώχευση είναι όλο και μεγαλύτερος. Είναι δύσκολο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των χωρών και να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο. Ποια είναι λοιπόν η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η λύση που προτείνουμε στη δική μας έκθεση, στην έκθεση IGS. Για να βγούμε από αυτή τη λογική, από αυτό το φαύλο κύκλο, θα πρέπει να βγούμε από αυτή τη φάση των υψηλών πολλαπλασιαστών. Θα πρέπει να μειωθεί η ανεργία, θα πρέπει να έχουμε σχεδόν πλήρη απασχόληση ή τουλάχιστον να, έχουμε, να βρεθούμε σε φάση μείωσης της ανεργίας. Σε μια οικονομία που έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης. Τότε η εμπιστοσύνη των οικονομικών φορέων είναι τέτοια που μπορεί αυτή η χώρα να έχει πρόσβαση στις ε, χρηματαγορές. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να έχουμε κάποια λιτότητα χωρίς να μειωθεί η οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει το έλλειμμα και το χρέος. Αντί δηλαδή να έχουμε υπερβολικά ψηλού στόχου για το χρέο και το έλλειμμα, βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να έχουμε πιο μετριασμένου στόχου, θα πρέπει να έχουμε μασοπρόθεσμους στόχου μείωση του ελλείμματο και του χρέου. Εύκολα το λέμε βέβαια αυτό, αλλά τίθεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν αναγγέλλεται ότι θα μειώσετε το μεσοπρόθεσμα, το χρέο και το έλλειμμα, πολλοί θα καταλάβουν ότι δεν θέλετε να το μειώσετε και ότι είναι ένα τρόπο να ξεφύγετε από τη λιτότητα θα κρατήσετε ψηλό το χρέο σα και τελικά θα δείξετε αμέλεια και δεν πρόκειται να περάσετε στην δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτός είναι ένας κίνδυνος και πρέπει να απαντήσετε σε αυτόν. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σύστημα όμως γι' αυτό όπου τα κράτη δεσμεύονται σε μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα. Και ποια είναι η λύση για να γίνει αυτό το πόμα. Για να έχουμε όλοι ξεκάθαρα, ξεκάθαρες ιδέες θα πρέπει για τα δημοσιονομικά θέματα να γίνει μια μεταφορά κυριαρχίας από τις χώρες προς τα νόμιμα θεσμικά όργανα για να αναλάβουν αυτή την κυριαρχία. Δεν είναι ούτε του Δουνουτού αυτό, αυτό το όργανο. Θα πρέπει να είναι αυτοί οι φορείς αντιπροσωπευτικοί, δημοκρατικοί, να μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση και να δουν τι πρέπει να γίνει. Αν περάσουμε σε αυτή τη μεταφορά κυριαρχίας, τότε μπορούμε να φανταστούμε μια άλλη πορεία για την ανάπτυξη πέρα από τη λιτότητα που θα επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε τα δημοσιονομικά, που θα επιτρέψει να φέρουμε το δημόσιο χρέος περίπου στο 20% να φύγουμε από την παγίδα της λιτότητας χωρίς όμως να διακινδυνεύσουμε μια κοινωνική ρήξη, οικονομική ρήξη, πολιτική ρήξη, κίνδυνο που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες και βεβαίως οι χώρες Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλοί είναι οι ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα τους ακούσουμε είτε με τη σειρά που υπέβαλαν το αίτημά τους, είτε με τη σειρά που τους είδα από την Bundestag της Γερμανίας, ο κύριος Μπάις, ο κύριος Λίντα, από την Επιτροπή Οικονομίας και Τεχνολογίας. Äh, Ευχαριστώ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή που προκαλεί πολλά ερωτήματα για την ανάλυση των ε, αιτίων της κρίσης και επίσης ε, για τις αντιφάσεις που εξεφράστηκαν. Στην ομιλία μου θέλω, μιλώντας κάπως ε, υπερβολικά, ότι δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο, δηλαδή από τη μία δημοσιονομική πειθαρχία από τη μία μεριά και από την άλλη μία οικονομική πολιτική που στοχεύει στη δημιουργία με τον ΑΒ τρόπο οικονομικών ε, προοπτικών για τις χώρες που έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Δεν είναι θέμα είτε. Είτε είναι και το μεν και το δε. Πρέπει να είναι σαφές ότι τι σημαίνει η φερεγγιότητα της χώρας, πώς μειώνονται, πώς μειώνονται το χρέος. Για όλα αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με το εάν η χώρα είναι σε θέση να συλλέξει τα έσοδα που χρειάζεται, αλλά και με τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της χώρας και τις προοπτικές συγκεκριμένα ανταγωνιστικότητας. Συμφωνώ κύριε Ζήν, αυτό αφορά το επίπεδο τιμών και μισθών, αλλά επίσης αφορά και τις ε, οικονομικές δομές, ε, τα κεντρικά σημεία της οικονομίας μιας χώρας και εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά στον τομέα της κατάρτισης, της έρευνας και στον τρόπο με τον οποίο μια χώρα μπορεί να διαφοροποιήσει την οικονομία της γύρω από τις διαπραγματεύσεις για, τη για το Διεσομικό Σύμφωνο έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα, αλλά πιστεύω ότι ακόμη περισσότερα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε οι χώρες που πλήττονται από την κρίση να έχουν μπροστά τους προοπτικές. Και μια τελευταία παρατήρηση. Κύριε Ζήν, αναφέρατε ότι παρόμοιες μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που έκανε η Γερμανία με το θεματολόγιο 2010 θα έπρεπε να ληφθούν και σε άλλες χώρες. Αυτό το συμμερίζομαι μόνο εν μέρη, γιατί δεν είμαι σίγουρος εάν παρόμοιες ε, μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα. Η Γερμανία είναι μια χώρα με καινοτομία, με ισχυρή βιομηχανική φάση, βάση. Έχει λοιπόν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό δεν ισχύει για όλους. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει περισσότερο συντονισμός και περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Ελλάδα τώρα, ο Αντώνης Μπέζας, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Πρόεδρε, Ζήτησα να μιλήσω σε αυτή την ενότητα τη ε, συνεδρίασης, όμω δεν μπορώ να μην κάνω μία αναφορά σε κάτι το οποίο υπόθηκε στην προηγούμενη ενότητα ε, στο πάνελ των ομιλητών. Άκουσα λοιπόν στην προηγούμενη ενότητα ότι από τον κύριο Κολινιόν, από τον καθηγητή Κολινιόν, ότι οι αποφάσει τη κυβέρνηση Καραμαλή, τη ελληνική κυβέρνηση εκείνη τη περίοδου, αναφέρομαι στην περίοδο 2007, 2008 και 2009, δημιούργησαν προβλήματα στην Ευρώπη και στου πολίτε τη Ευρώπη. Θα μου επιτρέψετε να πω μια και η Ελλάδα είναι ένα αγαπημένο αρνητικό παράδειγμα για πολλού, όπω για παράδειγμα για τον κύριο Ζην, ότι αυτή η άποψη, αυτή η προσέγγιση είναι εξαιρετικά απλοϊκή και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκείνη τη περίοδου έκαναν αποδεκτέ τι αποφάσει τη ελληνική κυβέρνηση και γενικά των κυβερνήσεων εκείνη τη περίοδου. Άρα, πού βρίσκεται το πρόβλημα το πρόβλημα βρίσκεται ότι στην οικονομική και νομισματική ένωση υπάρχουν συστημικές αδυναμίες και η κρίση η οποία δεν ήρθε ούτε από την ελλάδα ούτε από την πορτογαλία ούτε από την ισπανία έχει αναδείξει αυτές τις συστημικές αδυναμίες και την ανάγκη για την ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση και για ένα καλύτερο συντονισμό των πολιτικών σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης συντονισμός ο οποίος δεν υπήρξε στο πρώτο στάδιο της ελληνικής κρίσης. το ευρωπαϊκό Εξάμενο ορίζει το πλαίσιο για ένα πιο ολοκληρωμένο δημοσιονομικό συντονισμό λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών. αν και το ευρωπαϊκό εξάμεινο έχει μέχρι σήμερα μια επιτυχή θα έλεγα εφαρμογή πιστεύουμε ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω βελτίωση βελτίωση μπορεί να υπάρξει ιδιαίτερα στου τομεί τη δημοκρατική νομοποίηση υπόθηκε αυτό και από πολλού άλλου συναδέλφου προηγουμένω του καλύτερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και του συστήματο ελέγχου και λογοδοσία λογοδοσία τόσο στο επίπεδο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου όσο και στο επίπεδο των εθνικών κοινοβουλίων και σε αυτό το πλαίσιο για παράδειγμα μια πρόταση είναι οι ειδικέ αναχώρα συστάσει να μπορούν να παρουσιάζονται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και από τι εθνικέ κυβερνήσει στα εθνικά κοινοβούλια ενδυναμώνοντα έτσι ε, τη νομιμότητα τη δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία. θέλω να κάνω και άλλη μια ε, πολύ συγκεκριμένη παρατήρηση. Η έκθεση για το μηχανισμό επαγρύπνησης για το 2013 δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ελληματικών και των πλεονασματικών χωρών. είναι γεγονός ότι τελευταία αρχίζουν να διαφαίνονται κάποια αποτελέσματα στις πολιτικές της Ένωσης, αποτελέσματα γιατί τα ελλείμματα μειώνονται, οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχωρούν και υπάρχουν δείγματα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ακόμα υπάρχουν ορισμένες σημαντικές, θα έλεγα, θεσμικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να ελοπιθούν, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εξυγίανσης των Τραπεζών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Ένωσης και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εγγύησης των Καταθέσεων Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε δύο πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι συνεχίζεται ακόμη ο φαύλος κύκλος της ύφεσης. Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής στην ύφεση ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές οι οποίες είχαν εκτιμηθεί αρχικά. Οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές ήταν τελικά πολύ μεγαλύτεροι. Το αναγνωρίζει αυτό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η δική μου χώρα η Ελλάδα θα βρίσκεται το 2013 για έκτη συνεχή χρονιά σε κατάσταση ύφεση, διότι οι προβλέψει δεν έλαβαν υπόψη τι ιδιαιτερότητε και τι ιδιαίτερε συνθήκε που επικρατούν σε κάθε χώρα. Το δεύτερο είναι ότι το χάσμα ανταγωνιστικότητα, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω, μεταξύ των ελληματικών και των πλεονασματικών χωρών εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης και κοινωνικής ρήξης επομένως θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος το οποίο αποτελεί και μία από τις βασικότερες αιτίες της κρίσης είναι ευθύνη όλων των κρατών μελών. πρέπει πράγματι να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό ανταγωνιστικότητας. όμως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να γίνει μέσω μόνο από την απότομη εσωτερική υποτίμηση Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, μόνο μέσα από την απότομη εσωτερική υποτίμηση, γιατί αυτή οδηγεί σε κοινωνική εξαθλίωση. Τι να την κάνω την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα όταν έχω ένα λαό ο οποίο είναι κοινωνικά εξαθλειωμένο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε και άλλου τρόπου και παράλληλα θα πρέπει να προωθηθούν άλλοι στόχοι όπω η ενδυνάμωση τη βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασία. Και μία αναφορά στον καθηγητή, τον κύριο Ζήν, ο οποίο εμέσω, πλην σαφώ όμω, έθεσε το ζήτημα. Ο ελληνικό λαό έχει κάνει το τελευταίο διάστημα τεράστιε για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ και θα παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Η επιτυχία της Ελλάδος θα είναι και μια επιτυχία της Ευρώπης. Και η αποτυχία της Ελλάδος, τυχόν αποτυχία της Ελλάδος, θα είναι μια αποτυχία για το κοινό ευρωπαϊκό μας όραμα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πάνω κάτω τον απαραίτητο χρόνο, αρκεί όμως να τηρήσετε το όριο των τριών λεπτών. Διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έμιλι Τούρινεν. Ευχαριστώ. Μιλάω εξ ονόματος ομάδας των Πρασίνων, πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Κάποιες ερωτήσεις για τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Παρουσιάσεις Ερωτήσεις προς τον κύριο Σιν καταρχάς, αλλά μπορείτε και οι υπόλοιποι να απαντήσετε προφανώς. Ήταν κάπως καταθλιπτικό να σας ακούει κανείς, γιατί θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατον τελικά να βγούμε από την κρίση που υπάρχει στην Ευρωζώνη εξαιτία του τεράστιου χάσματος ανταγωνιστικότητας και του μεγάλου χάσματος στις τιμές. Είπατε ουσιαστικά να αυξήσουμε τη ζήτηση στο βορρά και να αφήσουμε τι δυνάμει αγορά να το κάνουν αυτό. Εγώ προέρχομαι από τη Δανία, έχουμε μια σχετικά υγιή οικονομία, καλά δημόσια οικονομικά, είμαστε εκτό Ευρωζώνη, αλλά μολονότι έχουμε αρνητικό κόστο δανεισμού, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, δεν υπάρχουν ιδιωτικέ επενδύσει. Δεν υπάρχει ουσιαστική πραγματική εμπιστοσύνη προκειμένου να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και ουσιαστικά οι δυνάμει αγοράς αγορά δεν παίζουν το παιχνίδι στο οποίο αναφερθήκατε. Δεν πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να αυξηθεί καταρχά η εμπιστοσύνη στο αύριο μέσω τη αύξηση των δημοσίων δαπανών στι χώρε εκείνε τη Ευρώπη που το χρειάζονται περισσότερο, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Πολωνία, κάτω χώρες προκειμένου να καταφέρουμε ουσιαστικά μέσω των πολιτικών αυτών να αυξήσουμε τη ζήτηση και να αυξήσουμε την κατανάλωση και την απασχόληση, ενδεχομένω να αυξήσουμε και του μισθού στι βόρειε χώρε, πράγμα το οποίο εγώ θα έκρινα θετικό και για τι νότιε χώρε. Δεύτερον, πώς μπορούμε ουσιαστικά να αγνοούμε ως παράγοντα τους μισθούς για την περίφημη αυτή ευθυγράμμιση στην οποία αναφερθήκατε. Είπατε ότι δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν οι μισθοί στον Βορρά με ένα τεχνητό τρόπο, με έναν αφύσικο τρόπο. Είπατε δεν θα ήταν θετικό αυτό. Πώς μπορούμε όμως να διαγράψουμε τελικά την επιλογή αυτή εντελώς. Τρίτον, έχουμε όλες αυτές τις ανισορροπίες. Αναφερθήκαμε σε αυτές, έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο και έχουν επεκταθεί με τα χρόνια. Πώς μπορούμε όμως, πώς είχαμε τελικά ένα επιτυχές ευρώ, μια επιτυχή οικονομία στην Ευρωζώνη όλα αυτά τα χρόνια, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Οφείλεται αυτό στη θετική οικονομική ανάπτυξη, η κρίση τελικά ήταν η μόνη η οποία κατέδειξε τις τεράστιες αυτές αποκλήσεις και ανισορροπίες. Τελευταία ερώτηση. Στα πλαίσια της Νομισματικής Ένωσης υπάρχουν πολλές ε, ανισότητες, αλλά έχουμε και μια κεντρική τράπεζα, έχουμε μηχανισμούς ανακατανομής και διαχείρισης ε, του χρέους. Δεν πιστεύετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα αυτά για να βρούμε την περίφημη διέξοδο για την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Από την Πορτογαλία, Πάολα Μοντεπίντο, επικεφαλής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρωτοβολία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μέσο του προγράμματος ανάκαμψης. Και βλέπουμε ότι οι εξελίξεις στη δευτερογενή αγορά μας επιτρέπουν για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια να είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Συνεχίζεται σαφώς η κρίση, αλλά βλέπουμε ότι η πολιτική προσαρμογής και οι μεταρρυθμίσεις της χώρας μου θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο. Η μέση επιχείρηση στην Πορτογαλία, με την πάνω κάτω ίδια παραγωγικότητα και αριθμό προσωπικού, εφόσον βρίσκεται στη Λισαβόνα, θα πληρώσει υψηλότερα επιτόκια από αν βρισκόταν κάπου αλλού στη χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού. Γιατί η εταιρεία στην οποία αναφέρθηκαν βρισκόταν στη Γερμανία θα πλήρωνε πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Διεξάγεται λοιπόν αυτή τη στιγμή μια συζήτηση στην Πορτογαλία για αυτή την περίφημη θεσιακή σπήρα και την όλη ιδέα ότι τελικά η ύφεση οδηγεί στην ύφεση χωρίς να επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση Πορτογαλίας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ξανακερδίσει ένα πρώτερο επίπεδο ταγωνιστικότητα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει υποτίμηση. Αλλά δεν θα ήθελα να σα δώσω αριθμητικά δεδομένα αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να σα πω ότι τα στοιχεία που έχουμε από τα τέλη του 2007 μέχρι το 2012 είναι σχετικά αρνητικά. Δηλαδή τα μόνα θετικά δεδομένα που έχουμε πλέον είναι το 2012, από το ότι υπάρξουν εφαρμόζονται τα μέτρα λιτότητας. Είδαμε προφανώς κάποιες ε, μειώσεις όσον αφορά τους μισθούς είχαμε σημαντικές μειώσεις και για τους δημοσίους υπαλλήλου, αλλά και για άλλου εργαζόμενου στην Πορτογαλία, όσον αφορά τι αποδοχές του πάντα. Κάτι ακόμα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να συγκρίνουμε τα επίπεδα τιμών με την Τουρκία, για παράδειγμα, όπως είπατε. Χώρα της οποίας η ε, ισοτιμία αγοραστικής δύναμης βρίσκεται μακριά ουσιαστικά από τα επίπεδα τα οποία έχουμε σε άλλε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε σαφώ όμως συντονισμό. Χρειαζόμαστε κοινέ πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική λιτότητος. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ο απαραίτητο συντονισμός λοιπόν. Αν δείτε τα όσα λέγονται για την Τραπεζική Ένωση, ε, τότε θα πρέπει όλα αυτά να ισχύουν με τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε, τελικά σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συντονισμό για τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και ένα συντονισμό και τις πολιτικές που βρίσκονται υπό επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλάβετε τι εννοώ αν συγκρίνετε δύο χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε τι γίνεται στην Πορτογαλία και τι γίνεται στη Γερμανία. Είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει τελικά να βγει από την κρίση αυτή, μόλον ότι ακούγονται κάποιε αρνητικέ εκτιμήσει αυτή τη στιγμή. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επόμενο ομιλητή, Βιάν Κόγκ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σάρον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μας ομιλητές που τελικά οι αποκλίνουσες αναλύσεις αντιστοιχούν στις δικές μας συζητήσεις εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο ερωτήσεις, ερωτήσεις και προς τους δύο μάλλον ομιλητές. Κύριε Σιν, είστε πάρα πολύ γνωστός στη Γερμανία. Θεωρείτε ότι η σκέψη σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και πλούσια. Στην παρουσίαση που κάνατε, νομίζω ότι ουσιαστικά θα μπορούσε να κάνει κανείς τρεις κριτικές. Είπατε ότι για να αντιμετωπίσουμε το ασυμμετρικό αυτό σοκ αναφερθήκατε σε μια προσαρμογή που πρέπει να γίνει μέσω των τιμών και μέσω διαρθρωτικών αλλαγών. Δεν αναφερθήκατε όμως καθόλου σε δημοσιονομικές μεταφορές οι οποίες θα μπορούσαν ε, να γίνουν μέσω του κοινοτικού προπολογισμού και ιδίω αν θεσπίζαμε κάτι το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή, ένα προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Δεύτερον, περιγράψατε κάποιους μηχανισμούς, ιδίως για τη Γερμανία. Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν μόνο αν υπάρχει ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τιμών. Ξέρουμε όμως ότι στη Γερμανία η ανταγωνιστικότητα είναι κυρίως μια ανταγωνιστικότητα που δεν λαμβάνει υπόψη στο κόστος. Αν δούμε πραγματικά ποιες είναι επιπτώσεις από τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, συνειδητοποιούμε ότι οι τιμές των εξαγωγών των γερμανικών δεν μειώθηκαν και ουσιαστικά αυξήθηκαν τα περιθώρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή 2% παραπάνω από την αγορά. Επομένως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν αφαιρθήκατε ακόμα από τη γαλλική αγορά, με συγχωρείτε, με 2% πάνω. Δεν αφαιρθήκατε στο σημείο αυτό. Μια τρίτη παρατήρηση. Μας λέτε ότι η οικονομία δεν περιορίζεται από την ζήτηση. Μπορούμε να το πούμε αυτό πραγματικά. Τη στιγμή που η χρησιμοποίηση της δυνατότητας παραγωγής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται 10% κάτω από το φυσιολογικό τους επίπεδο. Και προς τον κύριο Ταμπό κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, Ποια είναι η αξία που έχει σήμερα ο πολλαπλασιαστής ο δημοσιονομικός. Είπατε ότι έχετε κάνει κάποιους υπολογισμούς τελευταίους και πότε πιστεύετε ότι πραγματικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις επιπτώσεις της ανάκαμψης. Στην Γαλλία λέμε ότι το 2014 θα έχουμε μία ανάκαμψη. Ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι αξιόπιστη πληροφορία. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ η Πολωνική Γερουσία τώρα. Μάρεκ Ζουλοκόφσκι. Ευχαριστώ που είπατε το όνομά μου σχεδόν ολόσωστα. Καταρχάς συγχαίρω τους ομιλητές και από, τις ε, δύο, από τα δύο τμήματα της συζήτησης. Πρώτη ερώτηση προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τίθεται το ερώτημα, είναι δυνατή η ανάπτυξη χωρίς ε, λιτότητα ή είναι αναγκαία η λιτότητα. Άκουσα τα επιχειρήματα. Άκουσα χθες ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη χωρίς λιτότητα, ενώ η άλλη πλευρά θεωρεί ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα η λιτότητα. Ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, πολύ επίκαιρη είναι η ερώτηση που τέθηκε τι γίνεται με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης χωρί λιτότητα. Ξέρω ότι κάποια στοιχεία έχουν αποφασιστεί 11 χώρε, αποφάσισαν να τον εισαγάγουν. Θα είναι τμήμα των ιδίων πόρων του προπολογισμού της Ένωσης, θα πάει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και Έχουν εξαχθεί διδάγματα από την Σουηδική περίπτωση που δεν κατέληξε πολύ θετικά και η Σουηδία δεν είναι μεταξύ των χωρών που αποδέχονται αυτόν τον φόρο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η παρούσα ευρωπαϊκή κρίση σημαίνει ότι κάποιες χώρες πρέπει να κάνουν θυσίες και να υπάρχει κάποια μίνιμουμ συνένεση του λαού σε αυτά. Ερωτώ λοιπόν κάποια στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ιδιαίτερα οι συγκεκριμένες αναχώρα συστάσεις μπορούν να βοηθήσουν αυτό το τόσο σημαντικό και δύσκολο καθήκον. Να είναι δηλαδή ένα σημαντικό στοιχείο της εθνικής Για το ορισμένε φορές είναι καλύτερα να σταλεί κάποιο κάποιος απ' έξω ότι κάποιες θυσίες πρέπει να γίνουν. Η Πολωνία έχει προτείνει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση να επιτρέψουν, όπως είπε ένας Σουηδός συνάδελφος, στους ευρωβουλευτές να εισέλθουν στις εθνικές συζητήσεις, να αναφέρουν όλα τα επιχειρήματα, τεχνικά, κοινωνικά, ούτως ώστε να επηρεάσουν θετικά την κοινή γνώμη σε κάθε χώρα. Αλλά τώρα μία επιφύλαξη. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο καθήκον. Πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε τα δύο είδη επιχειρημάτων. Θα ήταν θαυμάσιο λοιπόν να υπάρχει μία διαδικασία επικοδομητική, ανοιχτή, δημοκρατική, χρονικά περιορισμένη. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε οι συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να γίνουν τελετουργικές, να γίνουν ρουτίνα να είναι απλώς ένα καθήκον που θα το κάνουμε τυπικά. Πρέπει να γίνει ουσιαστική λοιπόν συζήτηση. Αλλά στην πράξη κρίνεται η αλήθεια. Θα ήθελα λοιπόν οι συστάσεις για κάποιες χώρες να γίνουν δεκτές από τα εθνικά κοινοβούλια και να έχουν θετικά αποτελέσματα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε απτή απόδειξη ότι θα έχουμε απτά θετικά αποτελέσματα. Ο Μάρεκ είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Οικονομίας. Αλλά με συγκίνησε τόσο πολύ που είπα σχεδόν ολόσωστα το όνομά του που ξέχασα να πω το αξίωμά του. Πορτογαλία λοιπόν τώρα. Εντουάρδο Καμπίτο, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη σήμερα έχει καταδειχθεί η σημασία του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, του αποτελεσματικού συντονισμού, όχι όπως τα τελευταία δύο χρόνια, όπου γίνεται μια ε, ανταλλαγή κατηγοριών για το ποιος φταίει για την κρίση. Οι εξελίξεις τα τελευταία τρία χρόνια κατέδειξαν ότι ο οικονομικός συντονισμός είναι θεμελιώδους σημασίας αν θέλουμε η Ευρώπη να ξεφύγει από την κρίση. Και θα το επιτύχουμε μόνο εάν εργαστούμε από κοινού για την ε, διατήρηση του ευρώ. Νομίζω ότι όπως είπε και ο καθηγητής Ζιν, ε, είναι λυπηρό το ότι στο παρελθόν είχαμε ανταγωνιστικές προσπάθειες για να κατοχυρώσει ο καθένας την οικονομία του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να αποδεχθούμε μεθόδους που ε, λειτουργούν μόνο σε επιστημονικές θεωρητικές καταστάσεις ή σε δικτατορίες. Δεν πρέπει να θέτουμε το δίλημα μεταξύ λιτότητας ή οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και στρατηγική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δυνατότητα ως Ευρώπη ως ε, μια αγορά 500 ε, εκατομμυρίων καταναλωτών να καταδείξουμε την ανταγωνιστικότητά μας στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Τα στοιχεία που έχουν ε, δημοσιευθεί καταδεικνύουν ότι 12 από 17 της ζώνης ευρώ δεν είναι οικονομίες τύπου νότου, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν ε, διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος ή χρέους. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η κύρια οικονομία εκτός της ζώνης ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης ε, παραβαίνει τους κανόνες για το έλλειμμα και βλέπουμε ότι η στρατηγική τα τελευταία τρία χρόνια οδήγησε την Ευρώπη σε ύφεση και το 2013. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι η πορτογαλική εμπειρία καταδεικνύει ότι ήταν λάθος συνταγή. Θετικά αποτελέσματα που έχουμε τους τελευταίους μήνες στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία προκύπτουν λόγω κυρίως της παρέμβασης έστω και καθυστερημένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που συμβαίνει στην Πορτογαλία είναι σαφές παράδειγμα ότι εάν εφαρμόσουμε την πολιτική των προσαρμογών με απόλυτη ακαμψία έχουμε έκρηξη της ανεργίας, συνέχιση της ύφεσης γεγονότα δηλαδή που ποτέ δεν τα είχαμε σε περίοδο δημοκρατίας και το έλλειμμα διατηρείται σε επίπεδα που δεν είναι χρηματοδοτήσιμα, δεν είναι βιώσιμα. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες είναι ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους για όλους, μέσω πρόθεσμους, έχοντας συνείδηση ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς όλες αυτές τις χώρες που ανέφερα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα και Γερμανία. Άρα χρειάζεται ευρύτερη μεσοπρόθεσμη συνένεση, ευρύτερη από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Άννη Ποδηματά. Uh, uh, Ευχαριστώ τους ομιλητές, Σάρων, για τις θαυμάσιες παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να εστιαστώ στο θέμα της σύγκλησης. Παρά τις διαφορές ε, που είχατε στις απόψεις σας, παρόλα αυτά υπήρξαν και κάποια σημεία σύγκλησης στις απόψεις των δύο μιλητών. Θεωρώ ότι και οι δυο σας αξιολογείτε τα προγράμματα προσαρμογής που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη-μέλη. Όχι μόνο εκείνα που είναι υποκαθεστώς προγράμματος και μνημονίου, όπως η Ισπανία. Πιστεύω όμως ότι η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων δεν είναι θετική και στους δυο σας. Είπατε ότι Αναφερθήκατε μάλλον στη Γερμανία και καταλαβαίνω ότι έχετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο και το ρυθμό της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Σας θέτω λοιπόν το εξής ερώτημα. Αυτά τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής μπορούν να προσαρμόσουν τον ρυθμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ή θα πρέπει να δεχθούμε την ιδέα ότι σε αυτά τα κράτη-μέλη μια γενιά θα πάει χαμένη. Γιατί ο ρυθμός ανεργίας μαζί με την τεράστια μετανάστευση, μαζί με την εγκατάλειψη των ανθρώπων που έχουν φοβερά προσόντα και που μεταναστεύουν, ε, όλα αυτά δημιουργούν μια χαμένη γενιά σε αυτές τις χώρες. Αυτή η χαμένη γενιά και η αύξηση των ισοτήτων μεταξύ των χωρών μελών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τιμπό, αναφερθήκατε για την κοινωνική ρήξη, την οικονομική ρήξη, την πολιτική ρήξη. Μιλήσατε για τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στην ε, παιδεία και στις υποδομές. Πολλές χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε αυτούς τους τομείς. Η ποιότητα της ε, παιδείας, τι υποδομέ έχουν, τι περιβαλλοντική προστασία έχουν. Συνολικά νομίζω όλα αυτά επανέρχονται υπό το ερώτημα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωζώνης, συνολικά. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας επ' αυτού. Ο τελευταίος ομιλητής είναι από το Ισπανικό Κογκρέσο. Γκαμπριέλ Λορεάγα, νομίζω ότι το λέω καλά, ε, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης. Πολύ καλά προφέρατε το όνομά μου. Είμαι από την Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα για να διευκρινίσω κάποια στοιχεία που αναφέρθηκαν και σύντομα σχόλια. Πρώτον, η εξέλιξη του προπολογισμού στην Ισπανία για το 2012. Η δημοσιονομική εξέλιξη. Ξέρετε ότι ξέρουμε ήδη τα στοιχεία για το κλείσιμο του προπολογισμού, τα οποία είναι σχεδόν επακριβώς αυτά που είχαμε προβλέψει. Δεν υπάρχει καμία απόκληση στην εκτέλεση του προπολογισμού. Δεν ξέρουμε ακόμη τις δαπάνες, αλλά ξέρουμε ότι η εξέλιξη των δαπανών και αυτή μόνο μερικά δεκαδικά στοιχεία θα διαφέρει από τους στόχους. Αντίθετα λοιπόν από αυτό που υπόθηκε, τα στοιχεία του κλεισίματος του προπολογισμού του 12 θα καταδείξουν ότι ο ρυθμός που είχαμε δεσμευθεί να κάνουμε τις προσαρμογές τηρήθηκε. Έναντι αυτών των προσαρμογών που κάνουμε, η εξέλιξη του ΑΕΠ το 2012, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, είναι λίγο καλύτερο από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ίσως να έχουμε μία μείωση 1,3% ενώ η πρόβλεψη της κυβέρνησης ήταν για μείον 1,5% είναι πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις άλλων ε, διεθνών οργανισμών. Αυτή η πολιτική προσαρμογών λοιπόν δεν είχε ως αποτέλεσμα περισσότερη ύφεση από την προβλεπόμενη. Αυτό είναι σε αντίθεση με τις ε, μεγάλες οικονομίες της ζώνης ευρώ που σχεδόν όλες είναι σε ύφεση ενώ το τελευταίο εξάμεινο έχει σημειωθεί μία μικρή βελτίωση αυτή η εξέλιξη λοιπόν που πρέπει να την θεωρήσουμε καλή ή τουλάχιστον όχι τόσο κακή έχει να κάνει με την βελτίωση των εξαγωγών της Ισπανίας. Αυτό το στοιχείο λοιπόν ότι η Ισπανία είναι καθαρός εξαγωγέας έναντι των ε, μεγάλων οικονομίων της Ευρώπης, Γαλλία και Ισπανία καταδεικνύει την ανταγωνιστικότητά της, την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού τη κόσμου. Οι προσαρμογέ που γίνονται στην Ισπανία, με την τεράστια ανεργία βεβαίω, επιτρέπει να μειωθεί το κόστο εργασία με τρόπο τρομερό. Άρα βελτιώνονται ταχύτατα και οι εξαγωγέ. Άρα η εξωτερική ζήτηση μα βοηθάει στην ανάκαμψή μα. Πού οδηγούν όλα αυτά. Πιστεύω ότι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατές οι εσωτερικές προσαρμογές. Όταν υπάρχει βούληση να, να εφαρμοστούν ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τρόπο συνεπή, όταν υπάρχει επαρκής ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, όταν χρησιμοποιούμε σωστά τις υπάρχουσες πιστώσεις, η ανταπόκριση των οικονομικών ε, παραγόντων και των επιχειρηματιών είναι ταχεία. Βεβαίω το δράμα της ε, ισπανικής οικονομίας είναι το τεράστιο ποσοστό της ανεργίας. Η ανεργία βέβαια είναι αναπόφευκτη γιατί επιτρέπει ε, να περάσουν ανθρώπινοι πόροι από τους μη παραγωγικούς τομείς όπως οι κατασκευές σε άλλους τομείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή με ρυθμό ε, λογικά ταχύ. Σε αυτές τις συνθήκες αυτό που θα μας ε, βοηθούσε το λιγότερο θα ήταν η υπερβολική ακαμψία στα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί και να κάνουμε λάθος στους στόχους. Άκουσα τον καθηγητή Ζήν που είπε ότι αυτό που κάνουμε είναι μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του ευρώ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πριν δημιουργηθεί το ευρώ διότι οι οικονομίες του ευρώ έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχουν διαφορετικές εξελίξεις. Υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι, ασυμμετρικές συμπεριφορές κτλ. Και γι' αυτό υπάρχουν και πιο έντονα σοκ. Αλλά γι' αυτό ακριβώς όταν επιλέγουμε μια ενιαία οικονομία, ένα ενιαίο νόμισμα για τόση οικονομία, είναι επειδή θεωρούμε ότι οι μηχανισμοί εσωτερικής ελαστικότητας θα επιτρέψουν προσαρμογές. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να συγχύσουμε σε αυτή τη συγκυρία τους στόχους μας. Βεβαίως πρέπει να διατηρήσουμε πολιτική λιτότητας μέσω πρόθεσμα, αλλά να είμαστε πιο ευέλικτοι, ούτως ώστε οι προσαρμογές που θα γίνουν να βοηθήσουν τα θετικά στοιχεία που ήδη έχουν εμφανιστεί σε οικονομίες όπως της Ισπανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, η Μπετίνα Κούντλε από τη Γερμανική Βουλή. Ε, έχασα την κάρτα της, γι' αυτό δεν μπορούσα να πάρω το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι από την αρχή είχα δώσει την κάρτα μου για να μιλήσω στο δεύτερο τμήμα, γι' αυτό φαίνεται χάθηκε. Πρώτον, να υπογραμμίσω την πρόταση. Η λιτότητα και η ανάπτυξη δεν είναι αντιφατικές πολλά προγράμματα εξυγίανσης ε, σε διάφορους τομείς της οικονομίας καταδεικνύουν ότι χρειάζεται να μειωθούν οι δαπάνες σε διάφορους τομείς σε διάφορες ε, χώρες το πρόβλημα είναι ο υπερβολικός δημόσιος τομέας και όχι επαρκής ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Άρα είναι σκόπιμο ο δημόσιος τομέας να συρρυκνωθεί και να δοθούν κίνητρα για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις προτάσεις δηλαδή που θα κάνει. Οι προτάσεις της Κομισιόν ίσως προσανατολίζονται υπερβολικά σε καινοτομίες αντί να αναλύσουν τι μπορεί να ενισχυθεί σε διάφορες χώρες, τι μπορεί να καταργηθεί, τι προσκόμματα μπορούν να καταργηθούν για την ε, ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, καταπολέμηση της ανεργίας. Σίγουρα είναι ο κύριος στόχος μας αυτός. Αλλά πώς θα επιτευχθεί είναι το ερώτημα. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Να εισάγουμε εγγυήσει εγγυήσει θέσεων εργασία για τους νέους, για παράδειγμα. Αυτό δεν θα επέλυε το πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην εκλογική μου περιφέρεια έχουμε υψηλή προσφορά θέσεων ε, μαθητευομένων και δεν έχουμε πολλούς μετανάστες. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί μαθητές διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει επαρκής, επαρκές κίνητρο για τους νέους να κάνουν προσπάθεια να κατακτήσουν αυτές τις θέσεις μαθητευομένων. Γιατί έχουν υψηλές απαιτήσεις για το επίπεδο αποδοχών που θα πρέπει να έχουν. Επίσης, ε, οι πιστώσεις στον τραπεζικό τομέα. Σχετίζεται με την επιτήρηση των τραπεζών στη σημερινή συζήτηση. Με ξένησε κάπως ότι οι έννοιες τραπεζική ένωση και επιτήρηση των τραπεζών δεν διαχωρίζονται σαφώς. Αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να υπάρχει επιτήρηση των τραπεζών στην Ευρώπη για τις τράπεζες που είναι συστημικά σημαντικές. Τραπεζική ένωση σημαίνει πολύ περισσότερα. Τραπεζική ένωση σημαίνει ενδεχομένως η κοινή χρήση των καταθέσεων. Αυτό ε, δεν μπορεί να το δεχθεί αυτή τη στιγμή το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Να κάνω δύο ερωτήσεις στον καθηγητή Ζιν. Μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τραπεζική επιτήρηση στην Ευρώπη. Πώς κρίνεται τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν τράπεζες στην οικονομία. Και δεύτερον, εξηγήσατε ότι σε ορισμένα κράτη είναι, ερω... είναι ασαφές εάν δεν υπάρχει μηχανισμός προσαρμογής των ισοτιμιών θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη. Είπατε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στην Ένωση για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα πίσω και ούτως ή άλλως ε, για να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις για το ευρώ χρειάζεται ομοφωνία. Άρα αυτό σημαίνει πως το ευρώ είναι, το ευρώ είναι μια ανεπίστρεπτη διαδικασία. Ευχαριστώ. Έχετε 2.000 ερωτήσει ο καθένας και πέντε λεφτά να απαντήσετε. Κάντε ό,τι μπορείτε, τι να πω. Ίσως θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε λιγάκι, να μας δώσουν διερμηνείς λίγο περισσότερο χρόνο. Παρότι μετά από τόσες ώρες και με τόσες γλώσσες που έχουν ακούσει και μεταφράσει, τους αξίζει λίγη ηρεμία και κάποιο διάλειμμα. Ε, αυτό που είπε ο τελευταίο ε, ομιλητής από την Ισπανία. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το ευρώ. Όμως πρέπει να σεβαστούμε την ε, συνθήκη του Μάστριχτ. Το ίδιο θέλω να πω και στον Ευρωβουλευτή. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε μεγάλες δημοσιονομικές μεταφορές... σε αυτή τη φάση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα έπρεπε να, να μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Να φτιάξουμε την πολιτική ένωση. να φτιάξουμε δηλαδή την, οι Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε τη συνθήκη. Δεν μπορούμε να ζητάμε οι υπηρεσίε που απορρέουν από μία συνθήκη, α, αν δεν την έχετε υπογράψει τη συνθήκη. Πρέπει να υπογράψετε πρώτα τη συνθήκη. Τώρα έχουμε το ευρώ και το ευρώ σημαίνει κάποια πράγματα. Ε, θέλετε να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με τη συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ε, για να γίνουν κάποια πράγματα θα πρέπει να περάσουμε σε μεγαλύτερη πολιτική ολοκλήρωση. Εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να περάσουμε στις ΗΠΑ. Κάποιος μίλησε για δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, όπως και να το πείτε, δεν θέλω να πάω εκεί. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια συνολική συνθήκη να περιλαμβάνει τα πάντα. Αλλιώ δεν γίνεται τίποτα. Οι τράπεζε, δύσκολο θέμα. Φυσικά θέλουμε ε, μια κοινή εποπτική αρχή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι η ΕΚΤ, γιατί είναι τμήμα του προβλήματο. Έδωσε σε νότιες τράπεζες πολλά κεφάλαια χωρίς εγγύησει και επομένω είναι όμοιρο αυτών των δανείων δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο θεσμικό όργανο, δεν είναι αμερόληπτη για να αποφασίσει πώ θα γίνει η διάσωση. Για την ακεφαλαίωση των τραπεζών υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία. Ε, χρησιμοποιούμε τα λεφτά τον, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση. Υπάρχει μια μεγάλη διαφωνία μεταξύ των οικονομολόγων. 500 ε, οικονομολόγοι στη χώρα μου διαφωνούν. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση όμω. Ε, η χαμένη γενιά για την οποία κάποιο μίλησε. Πολύ σημαντικό. Όντω υπάρχει μια τέτοια χαμένη γενιά. Γιατί? Γιατί η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ κακή για κάποιε χώρε και προέκυψε από αυτή τη φούσκα που ξεκίνησε από το 1995 μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση. Τώρα θα πρέπει να μειώσουμε τις τιμές. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ένα-δυο μιλητέ είπαν ας κάνουμε την α μεταρρύθμιση, την β μεταρρύθμιση, υποδομές κτλ. Εντάξει, κάντε τα. Αλλά μην πιστεύετε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσει θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα χωρίς μείωση των τιμών. Όχι, όλα περνάνε μέσω τη μείωση των τιμών. Αυτές οι μεταρρυθμίσει αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και με δεδομένους τους μισθούς πρέπει να μειώσετε τις Έτσι γίνεστε πιο ανταγωνιστικοί. Ε, χρειάζονται, είναι χρήσιμες Α, ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα κανάλια. Και με κάποιο μαγικό τρόπο να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότητα. Λυπάμαι. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσω αναπροσαρμογής των τιμών. Και όταν το καταλάβουμε, καταλαβαίνουμε και το πρόβλημα και τη ρίζα του προβλήματος. Τα κενσιακά μέτρα αύξησης της ζήτησης. Ωραία, δημιουργούμε ένα, μια καλή, ένα καλό αίσθημα στον ασθενή. Α, του δίνουμε ένα αλγητικό. Αλλά δεν είναι εκεί η λύση. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και οι τιμέ θα πρέπει να είναι αντίστοιχε με την ε, ποιότητα του προϊόντος. Όλα αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται στην ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Οποιαδήποτε οικονομία της αγοράς έτσι πρέπει να λειτουργεί. Έτσι παγιδεύτηκαν διάφορες χώρες με τέτοιες ε, ψευδείς ιδέες στην Νότια Ευρώπη. Το να κρατήσουμε όλε τι χώρες μέσα και την Ελλάδα. Είναι αμαρτία εναντίον του ελληνικού πληθυσμού. Θα δημιουργηθεί αυτή η χαμένη γενιά αν το κάνετε. Γιατί το κάνουμε. Όχι για τον πληθυσμό. Λόγω των κεφαλαγορών. Όλοι ξέρουν ότι όσο η Ελλάδα παραμένει μέσα, όσοι έχουν τα ελληνικά ομόλογα μπορούν να ξέρουν ότι θα αποπληρωθούν, ε, θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Κάθε χρόνο που μένει η Ελλάδα, οι επενδυτές είναι σίγουροι ότι θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Νομίζω ότι έχουμε πάρει όμοιρο, οι κεφαλαίγορες έχουν πάρει όμοιρο τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν καλές ε, ευκαιρίες, ε, προσωρινή αποχώρηση με δυνατότητα επιστροφής. Καλύτερο θα ήταν για τις ε, εισαγωγές, για να βοηθηθεί ο τραπεζικός τομέας κτλ. Αν γίνει μια προσωρινή διατεταγμένη έξοδος, αυτή είναι η καλύτερη στρατηγική για τον ελληνικό πληθυσμό. Παρά να επιβάλλουμε αυτή τη στασιμότητα που οδηγεί τη χώρα στα όρια του εμφυλίου πολέμου. Και θα το κάνει αυτό σίγουρα μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια. Ορισμένοι δοκιμάσουν και τα δύνατα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αμαρτία εναντίον του πληθυσμού τους. Ένα-δύο άλλα ερωτήματα ακούστηκαν. Πώ προήλθε αυτή η κατάσταση, αυτή η κρίση ε, στην Ευρώπη, Γιατί είχαμε πολλέ μετακινήσει κεφαλαίων. Κάτι που ήταν χρήσιμο για την ανάπτυξη στον Νότο. Απέκτησε μεγάλη ορμή, δημιουργήθηκε η φούσκα των ακινήτων. Είχαμε τη δυνατότητα να αυξηθούν οι τιμέ, αλλά το όλο πράγμα ξεπέρασε το σημείο ισορροπίας. Έπρεπε να είχαμε ε, εφαρμόσει τροχοπέδες ε, σε αυτές τις κινήσεις κεφαλαίων νωρίτερα. Αν το είχαμε κάνει, δεν θα είχε δημιουργηθεί αυτή η φούσκα και δεν θα είχε σπάσει. Πυροδοτήσαμε πολύ αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Προήλθε όλη αυτή η πυροδότηση από τις κεφαλαγορές. Αλλά αυτό είναι λάθος. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Δεν μπορούν. Είναι αναγκασμένοι να είναι προσεκτικοί. Ε, Ξαγρυπτούν τη νύχτα για τις επενδύσεις τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στην Ευρώπη δημιουργήσαμε τεχνητά αυτή την αίσθηση της ασφάλειας. Το κάναμε αυτό από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ευρώ και αυτό δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα, όλη αυτή την αστάτωση για τους μισθούς. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε υψηλότερου μισθού στη Γερμανία. Πρέπει να έχουμε πληθωρισμό στη Γερμανία. Δεν μπορούμε όμω να επιβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον πληθωρισμό. Αν αυξήσετε απλώ του μισθού, ουσιαστικά επεμβαίνετε στον τομέα τη προσφορά. Ξέρετε ότι ε, ένα οικονομολόγο ουσιαστικά αν μειώσει τελικά την απασχόληση. Αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς μέσω της αύξησης της ζήτησης. Και αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο αυτόματο, φυσιολογικά απόλυτα από τις αγορές. Γιατί οι αγορές ουσιαστικά θέλουν τώρα να επενδύσουν στη Βόρεια Ευρώπη. Τόσα πολλά χρόνια δεν το κάνανε αυτό, τώρα όμως οι αγορές επιθυμούν να επενδύσουν στις βόρειες αγορές, πράγμα το οποίο σημαίνει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, αύξηση των μισθών Στη Γερμανία μετά από 15 χρόνια μείωση των τιμών των κατοικιών βλέπουμε τώρα ότι οι τιμές αυτές αυξάνονται. Όλοι ουσιαστικά κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και σιγά σιγά οι γερμανικές εξαγωγές θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές που είναι σημαντικές όμως για την αυτιγράμμιση που θέλουμε και θα αυξηθούν οι εισαγωγές. Και από τις δύο πλευρές λοιπόν πρόκειται να μειωθεί το έλλειμμα τραχουσών συναλλαγών. Η αύξηση όμως των μισθών δεν μπορεί να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο και αυτόματα. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί κανείς να αυξήσει μισθούς ή να προκαλέσει την αύξηση των μισθών. Ξέρετε, ορισμένοι πολιτικοί δεν κατανοούν καθόλου πώς λειτουργούν τα πράγματα στην οικονομία. Η κυρία Λαγκάρτ λέει ότι πρέπει να αυξήσετε πάντα τους μισθούς προκειμένου να μειώσετε το χάσμα στο σωζύγιο τρεχουσών εισαναλγών. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος να λέει αναλγον θεωρω οτι κανει παρα πολυ τέτοιο σφάλει απολύτως και δεν νομίζω πραγματικά ότι είναι οικονομολόγος. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος, αλλά σημαντικός, ο κύριος Ταμπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο. Είναι πολύ επικίνδυνο στην οικονομία και ιδιαίτερα στην μακροοικονομία να βασιζόμαστε σε κάποιες μεταφορές. Κάποιοι χρησιμοποίησαν τη μεταφορά του ασθενού στον οποίο δίνουμε ένα παυσίπονο. Και ότι αυτό δεν πρόκειται βέβαια να θεραπεύσει την ασθένεια. Θα μπορούσε να πεις και κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να επιβάλλετε, για παράδειγμα, σε κάποιον να κάνει μία δίαιτα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση αυτή ο ασθενή ενδεχομένω να πεθάνει από την ίδια τη δίαιτα και όχι από την ασθενειά του την αρχική. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στο εξή τώρα. Στα μακροοικονομικά κάνουμε αναλύσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Σήμερα έχουμε όλο και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές είναι υψηλοί. Θεωρούμε ότι οι επιπτώσει του σήμερα για την Ευρωζώνη στο σύνολό τη είναι ανάμεσα στο 1,3 και το 1,6. Για ορισμένε χώρε, όπω για παράδειγμα για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, έχουν ξεπεράσει το 1,5, βρίσκονται στο 1,5 με 2 Ορισμένοι αναφέρθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε ορισμένε χώρες, ορισμένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μπορεί να έχουν ω αποτέλεσμα να αυξηθεί επί τρία, να αντιπρελασιαστεί ο πολλαπλασιαστή. Μίλησα με τον κύριο Μπούτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ρώτησα ποια είναι η στάση της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι για το σύνολο της Ευρωζώνης οι πολλαπλασιαστές βρίσκονται ανάμεσα στον 1,2 και 1,7. Αλλά ακόμα και τα ποσοστά αυτά είναι υψηλά. Όταν προχωρά κανείς σε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις με τέτοιους πολλαπλασιαστές προφανώς προκύπτει ύφεση. Έχουμε δεδομένα θετικά από την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ναι, αλλά παράλληλα αυξάνεται και η ανεργία. Και παράλληλα έχουμε και ύφεση και όχι ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια κέρδη στο μέτωπο τη ανταγωνιστικότητα υπάρχει μια σχετική αύξηση των εξαγωγών, αλλά εξακολουθούμε και έχουμε ύφεση. Πρέπει να θέσετε λοιπόν το ερώτημα αυτό και πρέπει να αποδεχθείτε όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε τα έμπρακτα για τους πολλαπλασιαστές. Και θεωρώ ότι η λιτότητα, η δημοσιονομική λιτότητα ευθύνεται για την κατάσταση αυτή. Και θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Ενδεχομένως να έχουμε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες προκειμένου να δοθούν κάποια κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αληθεύει μεν αυτό, αλλά δεν μπορεί να το λέτε αυτό. Δεν μπορεί να λέτε ότι μπορείτε να έχετε μια λειτουργούσα οικονομία με μηδέν κράτος. Χρειάζεστε παιδεία, χρειάζεστε έρευνα, χρειάζεστε δημόσιες υποδομές. Αυτές φοβάμαι ότι θα χαθούν την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να το έχετε αυτό κατά νου. Και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικέ λύσεις. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι εξισορροπείται, αντισταθμίζονται οι πολύ μεγάλες ανισότητες στην Ευρωζώνη οι ανισότητες στην απασχόληση ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία αλλάζουν τις τιμές των, την, το επίπεδο των τιμών. Και το 20% δεν είναι πάρα πολύ ως προς αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ακολουθήσουμε τις αρχές της οικονομετρικής, τα επόμενα 10 χρόνια το επίπεδο των τιμών θα αυξηθεί και θα μειωθεί και το χάσμα αυτών των τιμών. Επομένως όλη αυτή η ιστορία της ανταγωνιστικότητας τελικά θα λυθεί θα ήθελα όμω να πω το ακόλουθο. Η ανταγωνιστικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την αύξηση των τιμών ανά στη ζώνη, στα πλαίσια τη Ευρωζώνη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και εκτό Ευρωζώνη. Κανεί δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε ότι έχουμε μια οικονομική, μια τριπεζική κρίση στην Ευρώπη, μια κρίση κρατικών ομολόγων. Τι θα γίνει όμω με τι υπόλοιπε χώρε. Όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα που κερδίζει αυτή τη στιγμή η Ισπανία με την υψηλή ενεργεία ουσιαστικά θα χαθεί στο μέλλον. Επομένως, πώς μπορούν να αντισταθμιστούν τα πράγματα. Λέμε πολλές φορές, ε, αναφερόμαστε στην υποτίμηση του δολαρίου και ότι αυτό ουσιαστικά θα οδηγήσει σε μια αύξηση ανταγωνιστικότητας στι Ηνωμένε Πολιτείε. Για ποιο λόγο να μην μιλήσουμε όμω περισσότερο για το ίδιο το ευρώ, γιατί να μην μιλήσουμε και μια συγκεκριμένη πολιτική όσον αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία. Για ποιο λόγο αφήνουμε μόνο τι Ηνωμένε Πολιτείε πραγματικά να κάνουν τη σημαντική αυτή συζήτηση για την αγωνιστικότητα. Θεωρώ ότι αυτό είναι τρελό πραγματικά. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η συνεδρίασή μας. Ξέρετε ότι προβλέπετε την αντίπνο στις 7. Αν δεν ξέρετε πρέπει να πάτε ζητήστε οδηγίες. Να ευχαριστήσω τους δερμηνείς, λέει πρόεδρος. Δεν ξέρω πραγματικά προς πως τρεις διερμηνείς σαν καμπίνα κατάφεραν τελικά να καλύψουν όλες αυτές τις γλώσσες. Σας ευχαριστώ πάντως πολύ. Η πρόεδρος ευχαριστεί τους συμμετέχοντες.